Uh, Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτό το τελευταίο τμήμα της συνεδριάσεως της Επιτροπής Ήτρε ξεκινήσαμε αυτό το πρωί. Λυπάμαι που δεν ήμουν εδώ μαζί σας. Ήμουν, βλέπετε, στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Συνέδριο, στο Κογκρέσο αυτό, για δύο μέρες. Έχουμε σημαντικότατο σημείο μπροστά μας. Σαν Επιτροπή Ήτρε είμαστε υπεύθυνοι για έρευνα, για καινοτομία, μαζί με τους φορείς της πραγματικής οικονομίας στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από Γεωργία και Αλία. Όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι τομείς εμπίπτουν σε αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Άρα πρέπει να αισθανθούμε υπεύθυνοι ιδιαίτερα για την τεχνολογική καινοτομία αλλά και άλλες καινοτομίες διότι ξέρουμε ότι η καινοτομία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά εν γέννη είμαστε υπεύθυνοι σαν καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα. Στο μέλλον, λοιπόν, θα αποφασίσουμε για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon Ευρώπη μεγάλος ωραίο όνομα Ορίζον Ευρώπη άρα φτάνει μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα είναι ο ορίζον της καινοτομίας που έχουμε θέσει τώρα είμαστε το μέσο του ορίζοντος 2020 ε, με άλλα λόγια το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερους καλεσμένους, του πιο σημαντικούς φιλοξενούμενους όσον αφορά τι μας Ο Επίτροπος ο κ. Μέντερς δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μέντερ που έρχεται εδώ. Καλώ ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέμα μας είναι επιστήμη και καινοτομία. Ανοιχτά στον κόσμο. Και παγκόσμιες προκλήσεις. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας του ένατου προγράμματος πλαισίου. Ο Επίτροπος ο κ. Μέντας θα μας πει κάποια λόγια γι' αυτό. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με το τμήμα το αρμόδιο για την αξιολόγηση επιστήμης και τεχνολογίας, με το πάνελ ΣΤΟΑ, σε συνεργασία με τη ΣΤΟΑ. Πρώτος αντιπρόεδρος της ΣΤΟΑ, ο κύριος Πολ Ρούμπικ είναι εδώ, εκπροσωπεί τη ΣΤΟΑ. Ο κύριος Πολ Ρούμπικ πριν από κάποια χρόνια ήταν πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος της ΣΤΟΑ. Τώρα είναι πρώτος αντιπρόεδρος. Καλωσορίζω θερμά και τον ιδρυτή και πρόεδρο του του Φόρουμ για την Επιστήμη Τεχνολογία στην Κοινωνία, τον κύριο Κόι Όμι. Χαίρομαι που σας βλέπω. Έχουμε μαζί μας αντιπροσωπευτικά άτομα, τον κύριο Μέντας, τον κύριο Ρούμπικ και τον κύριο Κόι Όμι τιμή για την Επιτροπή Ήτρε που φιλοξενεί μια τέτοια εκδήλωση του επίπεδου σε συνεργασία με, το Φόρουμ STS στη καθημερινό έργο της η Επιτροπή Ήτρε έχει κοινούς στόχους με το Φόρουμ STS και οργανώνει άτυπες συνεδριάσεις προς επίλυση συγγνώμη, των προβλημάτων που απορρέουν από τις εφαρμογές τις επιστημονικές και τεχνολογικές. Και τρίτο, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες από την Επιτροπή μας και όλους τους συμβούλους, τους βοηθούς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Επίτροπος, ο κ. Μαΐτας, είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος. Είναι πολύ σημαντικός και πάντα χρειάζεται κάποιους συνεργάτες που έχουν έρθει μαζί του σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση της Επιτροπής Ήτρε να έρθετε σήμερα στην εκδήλωση και να περιγράψετε τη διεθνή συνεργασία στο νέο πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη. Να μας πείτε ποιο είναι το όραμά σας. Πάντα μας χαροποιεί η παρουσία σας στις συζητήσεις μας και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία τους επόμενους μήνες όσον αφορά το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα Ορίζον ε, Ευρώπη. Για πρώτη φορά διαβάζω κάτι από το χαρτί. Συνήθως το λέω από απ' έξω. Εντάξει, δεν κάνει διαφορά. Τα ίδια θα έλεγα. Έχουμε ένα τρίωρο σχεδόν στη διάθεσή μας. Έχουμε τρία πάνελ. Εναρκτήρια συνεδρίαση και δύο θεματικές συνεδριάσεις. Μετά από κάθε συνεδρίαση παρουσίαση θα έχουμε ερωταπαντήσεις για ένα 20 λεπτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Κόι Όμι, ιδιωτή και πρόεδρο του Φόρουμ STS, για να μας κάνει μια εναρκτήρια ομίλια. Ευχαριστώ. Εξοχότητες, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ σε αυτή τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου που συνδιοργανώνεται από το Φόρουμ SES, τη ΤΟΑ και την Επιτροπή Ήτρε υπό την Προεδρία του δόκτορα Γέρζη Μπούζεκ που συμμετέχει για πρώτη φορά. Αυτή η συνεδρίαση είναι η τρίτη διάσκεψη που διεξάγεται εδώ, στις Βρυξέλλες, μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο και χάρη στις προσπάθειες του Δ. Πόλη Ρούμπικ, οργανώσεων την εκδίωση, και πρόεδρος του, του φόρουμ αυτού για την επιστήμη και τεχνολογία, το φόρουμ STS όπως αποκαλείται, αυτό το φόρουμ ετησίως συνεδριάζει κάθε Οκτώβριο στο Κιώτο, στην Ιαπωνία. Σε αυτό το βήμα το φόρουμ αυτό έχει μεγάλη επιρροή, διότι μαζεύονται πολλοί επιφανείς εκπρόσωποι που συζητούν επιστήμη και τεχνολογία, ειδικοί διαφόρων τομέων, ε, συνεδριάζουν, ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με το μέλλον της ανθρωπότητας. Τώρα είναι το 15ο έτος και το φόρουμ αυτό ο κ. Σιντοάμπε, ο Ιάπων Πρωθυπουργό, είναι ο τιμητικός πρόεδρος ε, στην ετήσια συνεδρίαση στο Κιώτο είχαμε 1.400 συμμετέχοντες από 80 χώρες. 35 υπουργούς επιστήμης τεχνολογίας μεταξύ άλλων, 46 ε, Πριτάνης πανεπιστημίων. Πάνω από 120 ανώτερους επιχειρηματίες είχαμε, ανώτερα επιχειρηματικά στελέχη. Το κ. Charles Holiday, πρόεδρο της ΣΕΛ, Royal Dutch Shell, τον κύριο Σαντούκη Ακιμπάρα, πρόεδρος, που είναι πρόεδρο της Οικονομικής ε, Ομοσπονδίας Ιαπωνία. Ο κύριος Μακίναλ, πρόεδρος ενός άλλου φορέα που είναι εδώ μαζί μας. Και ο κύριο Ταχέση Ουσουγεμάντα, πρόεδρος της Toyota Motors. Να αναφέρω μερικούς μόνο από αυτούς που συμμετείχαν. Σημαντικό λοιπόν να έχουμε ευρύ φάσμα ανθρώπων που συζητούν αυτά τα θέματα, που επηρεάζουν την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Εν αυτή τη έννοια φρονώ ότι το φόρουμ αυτό μπορεί να συμβάλλει σημαντικά μέσω του παγκοσμίου δικτύου ηγετών, επικεφαλής επιστήμες, επιχειρήσεις και σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις στον πολιτικό τομέα. Στη διάσκεψη αυτή, σήμερα, θα δούμε ποιο είναι το ίχνος του προγράμματος Ορίζον Ευρώπη και του σχετικού προγράμματος αυτού για το μέλλον. Θα είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτό στον κόσμο και αφορά προγράμματα καινοτομία και επιστημονικά που εφαρμόζεται παγκόσμια κλίμακα με τέρους από όλο τον κόσμο. Σήμερα σας φέραμε ηγέτη του, από το φόρουμ του STS φέραμε διάφορους ε, υψηλά αισθάμενα στελέχη από το φόρουμ αυτό για να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμφέροντος και πιο σημαντικό ε, υψηλά στελέχη της Ιαπωνικής κυβερνήσεως είναι εδώ μαζί μας. Και αυτό δείχνει το πόση σημασία έχει το φόρουμ και πόση σημασία δίδουν στη συνεργασία με την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φόρουμ STS λοιπόν προσβλέπει σε νέες ευκαιρίες που προσφέρονται από το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι χάρη στο ευρύ δίκτυο και την ευρεία συμμετοχή από όλο τον κόσμο, το Forum STS είναι ο ιδεώδης χώρος, το ιδεώδες βήμα. Είναι σε ιδεώδη θέση να συμμετάσχει ενεργά. Αυτό το σημαντικό πρόγραμμα θα ωφελήσει την ανθρωπότητα και είμαι ευγνώμων για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ενώσης Προσβλέπω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα και σε καρποφόρα αποτελέσματα για την υλοποίηση του προγράμματος για επιστήμη και τεχνολογία και ανάπτυξη. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω κάτι. Είμαστε αφοσιωμένοι αυτή η διάσκεψη, να συνεχίζεται αυτή η διάσκεψη ψηλού επίπεδου κάθε χρόνο. Σας καλώ να συμμετέχετε, να έρθετε στο φόρουμ του STS και στο παγκόσμιο δίκτυο του STS φόρουμ και ελπίζω να δω πολύ περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες σε ηγετικά στελέχη από την επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτικό κόσμο στην ετήσια συνεδρίασή μας στο Κιώτο από 7 μέχρι 9 Οκτωβρίου φέτος. Σας ευχαριστώ. Σα uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγική αυτή παρέμβαση αλλά και για την ε, διοργάνωση του φόρουμ αυτού που για μας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το φόρουμ STS αλλά και το πάνελ ΣΤΟΑ για την αξιολόγηση των τεχνολογικών επιλογών και επιστημονικών επιλογών. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και για την ομιλία σας, κύριε καθηγητά. Προχωρούμε στο εναρκτήριο τμήμα της συνεδρίασης. Πρώτη συνεδρία λοιπόν του ένα το πρόγραμμα πλαίσιο για τον Ευρώπη και τη διεθνή συνεργασία. Βασικός ομιλητής ο Επίτροπος, ε, κύριος Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος Αρμόδιος για θέματα έρευνας επιστημών και καινοτομίας. Περιμένουμε την πρότασή σας ε, και περιμένουμε να μας πείτε εδώ λίγα παραπάνω πράγματα για έναν από το πιο βασικό πυλώνα της πρότασής σας. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ Πρόεδρε κύριε Μπούζε, χαίρομαι πάντα που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Ήτρε και νιώθω πάντα την υποστήριξή σας, αλλά η σημερινή μέρα είναι ακόμη πιο ξεχωριστή, διότι έχουμε πραγματικά μια εξέχουσα ομάδα ε, ανθρώπων μαζί μας. Πρόεδρε, κύριε Ζιμπούζε, ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Παύλο Ρούμπι, ο οποίος από την αρχή ε, μου είχατε πει ότι πρέπει να είστε εδώ και είμαι εδώ για να συναντήσω μέλη της Επιτροπής Ήτρε και άλλους βουλευτές. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Όμη, Πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά σας να εδώ στην Ευρώπη και είναι πολύ καλό να ακούμε τα σοφά λόγια που πάντοτε εκφέρετε και τον κύριο Γιώση, τον Πρωθυπουργό επίσης σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, ε, τον κύριο Φωμικά Ζουσάτο. Πρώτα απ' όλα όμως, αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ε, για τους φίλους μας ε, κυρίως πρώτα από την, Ισπανία, από την Ιαπωνία που ήρθαν εδώ. Αν τυχόν υπήρχε κάποια αμφιβολία στο μυαλό οδήποτε ε, που δεν ζει στην Ευρώπη ότι δεν βάζουμε την καινοτομία και την επιστήμη στο επίκεντρο ε, του θεματολογίου μας ε, ελπίζω ότι δεν θα αμφιβάλλουν πλέον μετά την πρόταση που καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τον προπολογισμό επιστήμης και καινοτομίας. 100 δις ευρώ για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ορίζον Ευρώπη, έτσι το ονομάσαμε. Και πραγματικά είναι κάτι μοναδικό και συμβολικό. Γιατί για πρώτη φορά η πρόταση αυτή είναι τριψήφια ε, τα νούμερα τα οποία ε, προτείνονται. 100 δις ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι γιατί το χρειαζόμαστε απλά, αλλά γιατί είναι και μία δήλωση προς άλλα μέρη του κόσμου για τη σημασία που εμείς αποδίδουμε στην επιστήμη και στην καινοτομία. Και σε καιρό ε, αναταραχών εμείς βλέπετε ότι αναβαθμίζουμε τις δεσμεύσεις μας, τις αυξάνουμε. Αυτό είναι σημαντικό. και καλό είναι να δούμε ίσως και τι έγινε και κατά το παρελθόν. Για να γυρίσουμε λίγο πίσω στο 2000 που ήταν 15 δις ε, τότε ο προπολογισμό του προγραμματός μας. Και τώρα έχουμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς ε, το Κοινοβούλιο και προς τις χώρες μέλη, αλλά και προς το Κοινοβούλιο, του ε, των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φυσικά Είμαστε ευτυχεί και με καλή διάθεση γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ προσωπικά ξέρω ότι έχω την υποστήριξη όσων κάθονται σε αυτήν την αίθουσα και αυτό το θεωρώ καταπληκτικό. Σίγουρα πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν και θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο ακριβώς γι' αυτό, για το ανοιχτό του πνεύμα που θέλησε να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε σκληρά τους επόμενους δύο μήνες για να γίνει αυτό εφικτό και κυρίως για να μπορέσουμε να έχουμε διάλογο με τις χώρες μέλη. Είμαι βέβαιος ότι θα έχω την υποστήριξή σα και ελπίζω να έχουμε την υποστήριξη και των χωρών μελών. Σας ευχαριστώ θερμά όλους λοιπόν. Όμως, ο λόγος της επιτυχίας του προγράμματος αυτού, ο λόγος της επιτυχίας ε, του Ορίζοντα 2020 και των ε, προγραμμάτων πλαισίου που προηγήθηκαν, αν το σκεφτεί κανεί, ε, γιατί ήμασταν επιτυχημένοι, ποιο ήταν ο λόγο ε, της επιτυχίας και που οδήγησε σε αυτή την πρόταση των 100 δις. Τι κάνει διαφορετικά τα πράγματα. Και νομίζω ότι ένα από αυτά που κάνουν διαφορετικά τα πράγματα είναι κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ αυτών ο καθηγητής Μπουργκινιό που κάθεται εδώ, είναι στο κρατήριο, γιατί το βασικό είναι το να είμαστε ανοιχτοί. Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο είναι ένα υπόδειγμα ανοιχτού πνεύματος προς τον κόσμο Ποιο είναι το συστατικό του ανοίγματο, του ανοιχτού πνεύματο, ακριβώ το σημερινό μα θέμα, η διεθνή συνεργασία. Αν κανεί σκεφτεί τι θα πει διεθνή συνεργασία, τι θα πει άνοιγμα, ανοιχτό πνεύμα, ε, πρέπει να σκεφτεί και πώ ξεκίνησαν όλα αυτά. Είμαι Πορτογάλο ε, στην καταγωγή. Γιατί ε, δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ αν δεν ήταν οι Ιάπωνε φίλοι ε, και αν δεν σκεφτόμουν το άνοιγμα, το ανοιχτό πνεύμα του 15ου-16ου αιώνα. Οι συμπατριώτες μου ήταν αυτοί που έφτασαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία και το 1603 ε, μάλιστα έφτιαξαν και το πρώτο, ε, το πρώτο γλωσσάρι, ε, το πρώτο λεξικό για τη συνεννόηση των δύο λαών. Νίπο Τζίσο λέγεται αυτό το λεξικό. Και αν το διαβάσει κανείς, αν το ανοίξει, πάει στις ρίζες, πάει στις απαρχές αυτής της συνεργασίας. Και τι τελικά προέκυψε. Αυτοί που έγραψαν αυτό το λεξικό το 1603 έδωσαν ε, πορτογαλικές λέξεις και ιαπωνικές λέξεις για όλους. Και τι βλέπουμε σχεδόν 500 χρόνια μετά, ότι πολλές λέξεις παραμένουν κοινέ μεταξύ των δύο γλωσσών είναι σαν να μιλάμε με τις ίδιες λέξεις. Κόπο, που σημαίνει ε, φλιτζάνι, καντέια, σαμπόν, η σάπο, το σαπούνι, το κάπα, ε, το πανοφόρ κτλ. λοιπά Σχεδόν ίδιες λέξεις. Διεθνή συνεργασία λοιπόν ακριβώς αυτό σημαίνει. και στη χώρα σας την Ιαπωνία άρχισε πάρα πολύ νωρίς αυτή η συνεργασία με μια μικρή χώρα, την Πορτογαλία που όμως τότε ανακάλυπτε τον κόσμο. Σήμερα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το ανοιχτό πνεύμα σε μια στιγμή που ο κόσμος φαίνεται να θέλει κάπως να ομφαλοσκοπεί και να μαζευτεί στο καβούκι του. Έχω δίπλα μου τον πρόεδρο Μπούζεκ. Και θυμάμαι ότι είχαμε ε, προωθήσει την ιδέα αυτού ε, της, ε, του ανοιχτού χώρου καινοτομία έρευνας επιστημών. Ήταν τεχνικό στην αρχή και μετά από τρία χρόνια πήρε πολιτικές διαστάσεις. Ο κόσμος όταν ακούει αυτά που λέμε τώρα δεν ε, τα καταλαβαίνει όπως θα τα καταλάβαινε παράδειγμα πριν τρία χρόνια. Θα έλεγε ε, αυτός κάνει μια πολιτική δήλωση, αλλά δεν έπρεπε να γίνονται τότε πολιτικές δηλώσεις. Το θέμα είναι τώρα πώς οργανώνουμε σήμερα τον κόσμο. Uh, really the problem. Δείτε τι προβλήματα έχουμε σήμερα. Παντού στον κόσμο υπάρχουν ε, κάποιοι που θέλουν να γυρίσουν στο παρελθόν, αλλά αυτό το παρελθόν δεν υπάρχει πια και πρέπει να σας πω ότι και ένα παρελθόν που δεν ήταν τόσο καλό όσο ήταν το μέλλον είναι κάτι που δεν πρόκειται να γίνει. Ε, ένα παρελθόν που θα είναι καλύτερο από το μέλλον είναι κάτι που δεν υπάρχει. Κάποιοι το νομίζουν. Για να γυρίσουμε στο 19ο αιώνα, τι είχε γίνει τότε. Υπήρχαν οι λεγόμενες κάθετες αυτοκρατορίες. και το βασικό χαρακτηριστικό τότε ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ των αυτοκρατοριών αυτών. Έπειτα στον 20ο αιώνα από τις ε, κάθετες αυτοκρατορίες πήγαμε στις οριζόντιες, στα οριζόντια αλληλεξαρτώμενα μεταξύ τους έθνη. Και γινόταν λόγος εθνικό γόητρο, πώς μπορεί κανείς να είναι καλύτερος από το γείτονά του κτλ. Και τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα σήμερα με οργανώσεις και φορείς που είχαν σχεδιαστεί ήδη από το 19ο αιώνα αλλά πλέον μιλάμε για παγκόσμια δίκτυα. Να δείτε τους κόμβους, ε, πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα. Καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει ένα παγκόσμιο δίκτυο, ο μόνος τρόπος να επηρεάσει τα πράγματα δεν είναι ανταγωνιζόμενος ένας τον άλλο. Ούτε αυτοκρατές ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ούτε για εθνικά γόητρα μιλάμε, αλλά αυτό που μετράει τώρα είναι πώς μπορεί κανείς να επηρεάσει τα πράγματα. Και αν βρίσκεται κάποιο σε ένα δίκτυο κόμβων, με τρεις τρόπους μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Ο πρώτος τρόπος είναι με το ακριβώς αυτό ανοιχτό πνεύμα. Το ξέρουν οι πληροφορικάροι. Το δεύτερο είναι το ταλέντο και το τρίτο είναι λεγγύη και ένα πολύ καλό επιστήμονας και φιλόσοφος Μπακ Πάνα τα λέει πάρα πολύ ωραία όταν λέει συγκεκριμένα ότι ουσιαστικά η συνδεσιμότητα και όχι η κυριαρχία είναι ο νέος τρόπος οργάνωσης των ανθρωπίνων όντων στον 21ο αιώνα. Επιστήμη λοιπόν. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Ευρωπαίοι. Στο Nature υπήρχε ένα άρθρο πρόσφατα για την επιστήμη, την ανοιχτή που δημιουργεί πιο ισχυρέ χώρε. Τι θα πει ανοιχτή επιστήμη, θα πει πόσοι επιστήμονε φιλοξενούνται από ξένες χώρες ε, στη χώρα μας, πόσοι επιστήμονες από τη χώρα μας πηγαίνουν σε μια ξένη χώρα. Αν τους ε, προσθέσουμε αυτούς τους δύο, τις δύο κατηγορίες, αυτό θα πει ότι είμαστε ανοιχτοί στην επιστήμη. Όσο πιο ανοιχτή είναι μια χώρα στην επιστήμη, στους επιστήμονες, τόσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής αντικτύπου της επιστήμης. Δεν σας μιλάω για συναισθήματα εδώ, ούτε έρχομαι εδώ να σας μιλήσω ως πολιτικός για να σας πω ναι πιστεύω στο άνοιγμα, στο ανοιχτό πνεύμα, σας λέω. Τα λένε ε, τα επιστημονικά άρθρα, ε, οι επιστημονικές επιθεωρήσεις ε, ότι υπάρχει μεγαλύτερο συντελεστής αντικτύπου σε χώρες που είναι ανοιχτέ στην επιστήμη 20% υψηλότερο τελική σχέτισης Και ο αντίκτυπος. Και αν δείτε ποιε είναι οι 15 καλύτερε χώρες, οι πιο ανοιχτέ. δύο είναι που δεν είναι ευρωπαϊκές μεταξύ των 15. Καιρός είναι λοιπόν ίσως οι Ευρωπαίοι που τόσο καιρό μέσα στην κρίση ένιωθαν αποδυναμωμένοι, απογοητευμένοι, ε, καταρακωμένοι, που δεν λειτουργούσε η Ευρώπη. Φυσικά και έπρεπε να λειτουργούν τα πράγματα και σίγουρα ε, κάποια δεν λειτουργούν καλά, αλλά πολλά λειτουργούν. Και ένα από αυτά που λειτουργούν καλά είναι η επιστήμη και γι' αυτό πρέπει να είμαστε υπέρ. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ταλέντο. Το ταλέντο με φέρνει στο παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενωτικό Συμβουλίου και στον καθηγητή Μπουργκινιόν που είναι εδώ μαζί μας σήμερα of the European Research Council. Um... Ναι, Βλέπετε ότι αυτή, αυτό το άνοιγμα ε, βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση. Το 20% των ε, όσων συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα τη Ένωση έρχονται από άλλε χώρε του κόσμου. Σε ένα ψηφιακό κόσμο, το άνοιγμα αυτό δεν γίνεται μόνο από κάτω προ τα πάνω, από πάνω προ τα κάτω, αλλά και από κάτω προ τα πάνω πρέπει να γίνεται. Αν το κατανοήσουμε αυτό, θα αφανιστούμε. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ανοιχτοί και σε άλλους παράγοντες που σήμερα είναι σημαντικοί. Τις προάλλες διηγούν μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ που αποφάσισε πέκανα δύο χρόνια ήταν που αποφάσισε Έδινε ένα μάθημα το κωδικό 101 και είπε θα το κάνω στο ίντερνετ. Όχι με βιβλία, όχι με συνδράματα. Σκέφτηκε όμως και κάτι καλύτερο. Την εξέταση και αυτή να την κάνει στο ίντερνετ διαδικτυακά. Μάλιστα, υπάρχει φαίνεται ένα πρόβλημα, τα λέω πολύ γρήγορα. Έχω ενθουσιαστεί, ε, με έχει συνεπάρει το θέμα. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα το ταλέντο. Πώς έλεγα λοιπόν αυτός ο καθηγητής από το Στάνφορντ αποφάσισε να παραδίδει το μάθημά του διαδικτυακά αλλά και τις εξετάσεις να τις δίνουν οι σπουδαστές ε, διαδικτυακά. Και είχε δεκάδες χιλιάδες ε, νεαρούς και νεαρές από πανεπιστήμια ανά τον κόσμο που παρακολούθησαν το μάθημα ε, στο ίντερνετ και προσπάθησαν μετά να δώσουν και τις εξετάσεις ε, στο διαδικτύο και να τις περάσουν. Και το ενδιαφέρον είναι αυτός που πήρε το μεγαλύτερο βαθμό δεν ήταν αυτός, αλλά αυτή. Ήταν ε, μια νεαρή κοπέλα από τη Λαχώρη του Πακιστάν, 15 ετών σε ένα από τα πρώτα τέτοια ε, μαθήματα ε, του Στάνφορντ ε, που ξέρετε πόσο δύσκολο να μπει κανείς στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ είναι το πιο δύσκολο πανεπιστήμιο στη ΣΥΠΑ. Εγώ μπήκα στο Χάρβαρντ. Φανταστείτε ότι όποιος είναι στο Χάρβαρντ κοιτάει το Στάνφορντ και λέει πόσο δύσκολο είναι. Φανταστείτε λοιπόν μια 15χρονη από τη Λαχώρη του Πακιστάν να παίρνει το μεγαλύτερο βαθμό στο Στάνφορντ. Αυτό έγινε χάρη σε αυτό το άνοιγμα που επέτρεψε να φτάσουμε σε αυτή την κοπέλα στο Λαχώρη. Αλλιώ δεν θα το είχαμε πετύχει μέσω του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματο. Και ποιοι ήταν ε, μεταξύ των 20 ε, καλύτερων, ούτε ένα δεν ήταν από το Στάνφορντ. άκρο αποκαλυπτικό και αυτό. Μπορεί να είναι αστείο πιο πολύ αυτό που λέω, ανέκδοτο, αλλά η σημασία του είναι ότι όταν κανείς είναι ανοιχτό και αυτό όμως το επιτρέπει η ψηφιακή τεχνολογία, όταν λοιπόν ανοίγουμε προς τα έξω, ε, το ταλέντο εκδημοκρατίζεται κατά κάποιο τρόπο και προσεγγίζουμε πρόσωπα, άτομα που δεν θα μπορούσαμε να τα προσεγγίσουμε διαφορετικά. Μπαίνει δηλαδή πολλοί κόσμος μέσα σε αυτό το σύστημα που δεν θα μπορούσε να μπει αλλιώς. το Horizon Europe Ευρώπη που θα είναι το επόμενο λοιπόν πρόγραμμα ακριβώς αυτό το ανοιχτό πνεύμα, αυτή η διεθνή συνεργασία θα είναι το βασικό σλόγγαν και ο κινητήριο μοχλός. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει άνοιγμα όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν περισσότερο σε όσους θέλουν να είναι μέρη του συστήματος με ένα πρόγραμμα που θα είναι κλειστό και θα περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη δεν θα αποδώσει. Πρέπει να ανοίξει. Και σε πολλές άλλες χώρες. Επομένω, η πρότασή μου θα καταθέσω στο Κοινοβούλιο και θα τη συζητήσω με τους ευρωβουλευτέ, είναι να πάμε ε, στο επόμενο επίπεδο τη διεθνή συνεργασία. Σήμερα έχουμε πολλές ενώσεις, πολλές οργανώσει, αλλά πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε αυτές τις οργανώσεις. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση και σε άλλες χώρες, να βοηθήσουμε και άλλους να έρθουν κοντά μας. Θέλουμε δηλαδή να συμμετάσχουν χώρες που θα είναι μαζί μας για άλλους λόγους. Κάποιες ε, για την αριστεία, κάποιες γιατί έχουν καλύτερους επιστήμονες, κάποιες γιατί θέλουν απλά να μπουν στο παιχνίδι. Αυτό θέλουν για το μέλλον. Θέλουμε να είμαστε πιο ανοιχτοί στους διάφορους τομείς του προγράμματος. Όπως είπαμε λοιπόν στην πρότασή μας, θα έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Ανοιχτή επιστήμη, Open Science. Ένα πρόγραμμα παγκόσμιων προκλήσεων, Global Challenges και ένα πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας, Open Innovation. Είναι φανταστικό που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, και συζητώ μαζί σας αυτό το θέμα. Αν υπάρχει ένα στοιχείο από το ορίζον Ευρώπη που μπορεί να μας κάνει διαφορετικούς εδώ στην Ευρώπη από άλλα μέρη του κόσμου, είναι ακριβώς αυτό το ανοιχτό πνεύμα, αυτό το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Uh, thank Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Έξοχες εξηγήσεις που δώσατε. Παρουσιάσατε έξοχα μία από τις βασικέ ιδέες του προγράμματος Πλαισίου 9 Παρουσιάσατε λοιπόν τη θέση σας, τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρουσίασή σας ήταν σαφέστατη. Ως συνήθως ευρεία προσέγγιση, φιλοσοφική προσέγγιση, απόλυτα αναγκαία, ούτω ώστε το πιο θεμελιώδες θέμα να τεθεί. Το σημείωσα. Πώς οργανώνουμε τον κόσμο σήμερα και το έργο μας σήμερα. Βαθύ ερώτημα. Και το πρόγραμμά μας θα μπορούσε να μας βοηθήσει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βρούμε έναν δρόμο σαν δύσκολο κόσμο σήμερα. Ανοιχτή προσέγγιση, ταλέντα, ε, πολύ σημαντικά θέματα για μας. Αν επιτρέπετε, να καλέσω το δεύτερο ομιλητή για μια σύντομη παρέμβαση. Σύντομες παρεμβάσεις παρακαλώ. Ο κ. Γιώηση Ήτο, υφυπουργός παιδείας, πολιτισμού Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας και έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας από τον Ιούλιο του 2017 ως υπουργό και η δραστηριότητά σας στο βιογραφικό είναι τεράστια, ατομική ενέργεια. Στην πρεσβεία σας στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαβίω, πολιτική διαβίω εκμάθησης στην υπηρεσία της Ιαπωνίας στην νομική ενέργεια, αξιολόγηση πολιτικής, ε, προσέγγιση αφορά την πολιτική της αποφάσεων. το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ αξιότιμε Ζέρζι Μπούζεκ, αξιότιμε κύριε Ρούμπικ, αξιότιμε κύριε Μόεδας και αξιότιμες κυρίες και κύριοι, λέγομαι Ιώση Ήτο του Υπουργείου Επιστημών, Τεχνολογίας κλπ. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που απευθύνω τον λόγο σε εκπροσώπους όλων των τομέων της κοινωνίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ενδιαφέρονται για θέματα τεχνολογίας και επιστήμης. Σε ό,τι αφορά το ένατο ερευνητικό πρόγραμμα που, εξήγησε μόλις ο Επίτροπος Μόελας, ακούω ότι ο προϋπολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά. Αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι είναι αποφασισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδίδει μεγάλη σημασία στην επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία. Ο Horizon Europe έχει δύο ή μάλλον τρεις καινοτομία, επιστήμη και ανταγωνιστικότητα. Οι τρεις αυτοί πυλώνες έχουν πολλά κοινά στοιχεία με την ιαπωνική πολιτική για την επιστήμη και την τεχνολογία. STI λέμε εμείς συντομογραφικά στα αγγλικά. Δεν υπάρχει ακόμα βέβαια ολόκληρη εικόνα του νέου σας προγράμματος, αλλά θα ήθελα να έρθουμε στην επόμενη πρωτοβουλία και τη συνεργασία μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τρεις πυλώνες του προγράμματος ερευνών. Σε ό,τι αφορά την Ιαπωνική προσπάθεια, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε την Ιαπωνία την πιο φιλική στην καινοτομία χώρα του κόσμου. Ο οργανισμός τεχνολογίας και καινοτομίας υπό την εποπτεία του Υπουργείου μου προωθεί δραστηριότητες καινοτομίας τεχνολογίας από την πιο βασική έρευνα μέχρι πρακτικές εφαρμογές και διάθεση στο εμπόριο με τρόπο συνεκτικό και διαρκή. Κάνουμε προσπάθειες να στηρίξουμε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, start-up των αποφύτων των πανεπιστημίων. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ESE, έχει παρόμοιο ρόλο με το δικό μας EST. Θεωρώ λοιπόν ότι το JST και το ESE, e, οι δύο φορείς, δηλαδή ευρωπαϊκός και ιαπωνικός, μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα τις παγκόσμιες προκλήσεις, η Ιαπωνία με το STI, Science Technology Innovation, ε, εγκύπτει και σε κοινωνικά θέματα. Θεωρούμε ότι η ιδέα της επίτευξης των στόχων Βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών του 2015 έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν και αποφασιστικό ρόλο θα είναι του STI για την επίτευξή τους. STI for SDGs δηλαδή, πάλι σε συντομογραφίε στα αγγλικά. Έχω πολλές, πολύ μεγάλες προσδοκίες από τη συνεργασία των ε, δύο φορέων ε, Ευρωπαϊκού και Ιαπωνικού για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Βεβαίως η βασική έρευνα είναι σημαντική γιατί είναι θεμελιώδης για όλες τις δραστηριότητες STI. Στηρίζω την ιδέα του Horizon Europe να στηρίξει δηλαδή με τη σειρά του την βασική έρευνα και την ανοιχτή επιστήμη ως ένα από τους βασικούς πυλώνες του. Θα ήθελα όμως να ρίξουμε μια ματιά και στις ανταλλαγές διεθνών επιστημόνων. Πάνω από 9.000 Ευρωπαίους ερευνητές, Ευρωπαίοι ερευνητές μάλλον, ήλθαν στην, έρχονται μάλλον κάθε χρόνο στην Ιαπωνία και το αντίθετο. Ε, έτσι λοιπόν είναι από 20 έως 30% των διεθνών ανταλλαγών μας επιστημόνων. Και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει σημαντική θέση ως προορισμός Ιαπωνών ερευνητών. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της σημερινής συνεδρίας Horizon Europe και Διεθνή Συνεργασία τον Ιανουάριο του 2018 ο υπουργό μα Χαγιάση συναντήθηκε με τον Επίτροπό σας Μοεντά για να συζητήσουν θέματα επιστημονικής τεχνολογίας, επιστημονικής μάλλον συνεργασίας. Ελπίζουμε ότι η συνεργασία στην έρευνα μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχίσει ομαλά. Θα χαρούμε πολύ αν το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα είναι να είναι ανοιχτό και σε ερευνητέ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση. Στις συζητήσει μεταξύ του Υπουργού μα και του Επιτρόπου σας συζητήσαμε για ειδικού τομείς, ανταλλαγέ νεαρών ερευνητών και έρευνα στην Αρκτική. Σε ό,τι αφορά τους τομείς αυτούς έρευνας, με χαρά μου σας λέω ότι η συγκεκριμένη προετοιμασία για κάθε ένα από τα θέματα αυτά προχωρεί. Ένα παράδειγμα για την κβαντική τεχνολογία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που προσεκλήθη η Ιαπωνική ερευνητική ομάδα στην προηγούμενη εβδομάδα στην Γερμανία στην ε, συνεδρίαση της ε, ε, Επιτροπής Κβαντικής Τεχνολογίας και θα σας προσκαλέσουμε και εμείς, θα προσκαλέσουμε τους ερευνητές αυτούς στην Ιαπωνία. Η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας υπογράφηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Είμαστε λοιπόν εταίροι που έχουμε πολλά κοινά σημεία. Η συνεργασία μας στην τεχνολογία γίνεται όλο και πιο σημαντική ως πυλώνας της συνεργασίας μας. Ελπίζω ότι το πρόγραμμα Rising Europe θα στηρίξει ακόμα περισσότερο την περαιτέρω εξέλιξη και ελπίζω ότι το σημερινό εργαστήριο θα αποδειχθεί καρποφόρο για όλες και όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, Παρόμοιο σχόλιο έχω. Ήσασταν λίγο γρήγορος, αλλά τα καταφέραμε. Τώρα, λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω για την ομιλία σας, κύριε Γιωήση Ήτο, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Σύντομη παρέμβαση τώρα του κυρίου Φουμικάζου Σάτο, υποδιευθυντή για βιομηχανική επιστήμη και τεχνολογία σχετική πολιτική και υπηρεσία για το περιβάλλον του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανία. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά υπουργεία στην Ιαπωνική κυβέρνηση και στο βιογραφικό σας βλέπω πολύ δραστήριο Επιτροπή για τα πρότυπα τα Ιαπωνικά το Προεδρείο των Κατασκευαστικών Βιομηχανιών, Υπουργό Διεθνού Εμπορίου και Βιομηχανία, ανήκετε και στην αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη χώρα σα και διευθυντή για, για το ε, τμήμα ευημερία, για τι νεοεφυεί επιχειρήσει, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πάρα πολλέ δραστηριότητε. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον για μα να σα ακούσουμε Κύριε Φουμικάζου Σάτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε του STS, εξοχότητά σας κύριε Σκάλος Μίδες, ε, Μέντες, Επίτροπη της Ευρωπαϊκής Ενώσης, με κύριε Ρούμπι και κύριε Μπούζεκ, διακεκριμένοι φιλοξενούμενοι, κυρίες και κύριοι, Είμαι ο Φουκουσίμα Σάτο, υπουργό από το Υπουργείο Οικονομία και Βιομηχανία τη Ιαπωνία. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμησή μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας έδωσε μια πολύ καλή ε, ευκαιρία να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση σήμερα που είναι μεγάλη ευκαιρία. Και είναι τιμή μου που σας απευθύνω το λόγο αυτό. Σήμερα θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο, η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Δεύτερο σημείο, η σημασία της ανοιχτής καινοτομία. Και τέλος η τρέχουσα πολιτική του Υπουργείου όσον αφορά την επιστήμη και τεχνολογία. Πρώτα απ' όλα, Έχουμε το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο και διεθνή συνεργασία σε βασικό θέμα. Η Επανία διεξάγει κοινή έρευνα και ανάπτυξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της βιομηχανικής τεχνολογίας. Παραδείγματο χάρη, ε, το Εθνικό Ινστιτούτο Προωθημένης Βιομηχανικής Επιστήμης και Τεχνολογίας συμμετέχει στο πρόγραμμα Στάσερ που αναπτύσσει προϊόντα για τη δημιουργία τεχνολογίας νέας γενιάς για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020. Οι ιαπωνικές εταιρείες και τα ερευνητικά Ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάστηκαν σε προγράμματα πολιτικής αεροπορίας. Για το Sunjet 2 μαζί συνεργαστήκαμε για να αναπτύξουμε ε, ελαφρύτερα μικρότερα συστήματα ελέγχου πτήσεως και προθυμένα συστήματα αεροσκαφών για αποτελεσματικό χειρισμό των αεροσκαφών και υλικά ελαφρά νέας γενιάς. Αυτά τα προγράμματα είναι παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας και αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Πιστεύω ότι είναι καλή πρακτική να δημιουργούνται νέες τεχνολογίες μέχρι κοινή έρευνα και ανάπτυξη μεταξύ Ιαπωνία και Ευρωπαϊκής Ενώσεω, εποφελούμενοι από τα ισχυρά σημεία του καθενό μας. Είναι εύκολο να έχουμε ε, επαφέ με τους φίλους μας Ευρωπαϊκής Ενώσεω και αυτό βοηθά. Δεύτερο σημείο. Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο εξετάζεται και θα διαδεχτεί το πρόγραμμα Horizon 2020. Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο έχει τον τίτλο Ορίζον Ευρώπη και περίπου 100 δις ευρώ θα διατεθούν για αυτό το σκοπό βάσει του σχεδίου προπολογισμού που ανακοινώθηκε στις 2 Μαΐου. Το Ορίζον Ευρώπη θα ξεκινήσει το 2021 και έχει σχεδιαστεί γύρω από τρεις πυλώνες ακολουθώντας τη βασική δομή του ορίζοντα 2020. Ο πρώτος πυλώνας είναι ανοιχτή επιστήμη Δεύτερος πυλώνας είναι οι παγκόσμιες προκλήσεις και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και ο τρίτος πυλώνας είναι η ανοιχτή καινοτομία. Αυτοί οι πυλώνες επίσης τονίζονται στην Ιαπωνία. Εμείς εστιαζόμαστε στην ανοιχτή καινοτομία, εξ λίας Αλίας Φερρυπίν. Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα μέσω ανοιχτής καινοτομία στην Ιαπωνία. Άκουσα τα πιλωτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία με σκοπό την εμπορευματικοποίηση καινοτόμων ε, ιδεών και την υποστήριξη επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων. Εμείς θα συνεργαστούμε στα πλαίσια του ορίζοντα Ευρώπη. Είναι πολύ επίκαιρη η προσέγγιση που ακολουθούμε Τρίτο σημείο. Να υπογραμμίσω ότι το ΜΙΤΙ ε, επίσης εφαρμόζει πολιτικές για να υποστηρίξει την ανοιχτή καινοτομία Φερρυπίν, εμπορευματοποίηση τη έρευνα και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστηρίζεται με συνεργασία με ερευνητικά Ινστιτούτα και παρέχουμε υποστήριξη στην αυξανόμενη συμμετοχή στα διάφορα εθνικά προγράμματα έρευνα και ανάπτυξη. Κάποια πανεπιστήμια από κοινού έχουν δημιουργήσει εργαστήρια ανοιχτή συνεργασία για να εμπορευματικοποιήσουν τεχνολογίε που έχουν στην κατοχή του τα πανεπιστήμια και τα διάφορα ερευνητικά ιδρύματα. Σαν αποτέλεσμα αυτού μπορούν να αναπτύξουν πρακτικές εφαρμογές μέσω κοινή έρευνας και ανάπτυξης που εξαρτάται τις ανάγκες των εταιριών. Πρώτα απ' όλα, δημιουργούμε εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης με ιδιωτικές εταιρείες για να γίνει μεταφορά τεχνολογίας από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά Ινστιτούτα προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τώρα θα ήθελα να συνοψίσω ότι η ανοιχτή καινοτομία είναι απαραίτητη για να ξεπεράσουμε τα παγκόσμια προβλήματα και με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και αγορών. Για να αναπτύξουμε καλύτερη μελλοντική κοινωνία που θα είναι ευημερή και οι απόγονοί μα να ζούσουν σε ευημερία, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία να μοιράζονται τα αποτελέσματα τη έρευνα και ανάπτυξη και μέσω αυτών των εξελίξεων και αναπτύξεων να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τα SDGs όπως αποκαλούμε από τα αρχικά τους, ε, βάσει προτεραιοτήτων που έχουμε καθορίσει. Υπάρχουν έξοχες εταιρείε και ερευνητικά ιδρύματα και στην Ιαπωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η κάθε πλευρά ε, θέλει να είναι συμπληρωματική προσέγγιση. Να ενισχύουμε τα σχερά μας σημεία, ημέν τον δε, μέσω τη συνεργασία μας και ανάπτυξη Ιαπωνία και Ευρωπαϊκή Ενώσεω, που να χρησιμοποιηθεί αυτή για να απειληθούν παγκόσμια προβλήματα, όπω η αλλαγή του κλίματο, και να πετύχουμε του στόχου ε, τη ε, αναπτύξεω. Θα είναι υποφελής για όλους αυτή η συνεργασία στα πλαίσια του ορίζοντα Ευρώπη. Ειλικρινά, Ελπίζω ότι το σημερινό εργαστήριο θα είναι ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Uh, thank you very... Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενική Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ και τους δύο. Ακούσαμε συγκεκριμένα παραδείγματα οργανώσεως της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα σας και της ανοιχτής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά ήταν πολύ καλά, πολύ ενδιαφέροντα για τις προοπτικές που έχουμε. Θα σας καλέσω τώρα να προβούμε σε μια σύντομη συζήτηση, να συμμετάσχει το κρατήριο. Κυρία μου, η κυρία Κουντέσκα είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις φυσικά προς τον Επίτροπο. Συμφωνώ κύριε Επίτροπε μαζί σας. Η επιστήμη είναι ισχυρό διπλωματικό εργαλείο. Έχοντας κατά νου την αύξηση του λαϊκισμού και τις όλο και πιο προφανούς ε, κρίσεις της δημοκρατίας σε διάφορες χώρες μέλη, μήπως θα πρέπει να ενισχύσουμε αντίθετα την ε, θέση των χωρών ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο. Για το Horizon Europe συμφωνώ αλλά θα πρέπει να είναι ανοιχτό και στις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις, το ίδιο και για τις περιφέρειες ε, με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Θα ακούσετε ε, και θα ακολουθήσετε τα όσα είπε ο καθηγητής Λαμή. Καναδάς, Αυστραλία δηλαδή θα συνδεθούν. Πώς αυτό θα επηρεάσει την υφιστάμενη ερευνητική συνεργασία και τα σχετικά μοτίβα Ποια είναι τα αναμενόμενα ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποιου τομεί θα συνεργάζεται με αυτέ τι χώρε η Ένωση, ειδικότερα Αυστραλία και Καναδά. Οι φορεί του ε, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το καθεστώ Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Βραζιλία ε, έχει αλλάξει ε, αρκετά. Διεθνή συνεργασία στον ορίζοντα 2020 θα ακολουθήσει τις συστάσεις ε, του κυρίου Λαμή για μια πιο κεντρική δομή και τέλος πιστεύω ότι πρέπει να εκπονήσουμε μια έκθεση για τα αναλυτικά αποτελέσματα της διεθνούς συνεργασίας μας με τρίτες χώρες. Πρέπει να χαρυπώ πόσες σημαντικές δημοσιεύσεις είχαμε, πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ε, πόσα ταλέντα έχει κερδίσει η Ευρώπη, σε πόσα ερευνητικά προγράμματα συμμετέχει η Ευρώπη. Αυτή η έκθεση θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό γιατί θα ενισχύσει την ανοιχτή αυτή προσέγγιση που θέλει να ακολουθήσει η Κομισιόν κατά την άποψή. Επίσης, η Κομισιόν θα αλλάξει τον ορισμό τρίτης ή συνδεδεμένης χώρας και τους όρους συμμετοχής τέτοιων χωρών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, έχοντας υπόψη τον Brexit, Λίγες μέρες ή εβδομάδες μάλλον πριν από την παρουσία του ορίζοντα Ευρώπη δεν ξέρω αν είναι νωρίς για να μας δώσετε μια ιδέα για το ποιο θα είναι το καθεστώς ε, της μετά το Brexit. Thank you very much. Εγώ θέλω μόνο να συγχαρώ τον ίδιο τον κύριο Επίτροπο, όχι μόνο για την σύνταξη του προϋπολογισμού που βρίσκω ότι είναι από τους πιο φιλόδοξους προϋπολογισμούς για το πρόγραμμα, δηλαδή για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και για την ιδέα που προβάλλει το κόνσεπτ, που είναι σημαντικό για την διεθνή συνεργασία. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συμπέρασμα της Midterm Review ζήτησε βελτιωμένη συνεργασία, βελτιωμένη διεθνή συνεργασία. Για μένα αυτό είναι κρίσιμη σημασία τρόπος εργασίας. Συγχαίρω επίσης και την Ιαπωνική πλευρά. Αντιλαμβάνομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία έχουν παρόμοια, βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση στην εξέλιξη και αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές και παγκόσμια. Το πιο ενδιαφέρον που άκουσα σήμερα είναι η συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, της, ε, των βιώσιμο, της βιώσιμης ανάπτυξης δηλαδή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, ποια θα είναι η σχέση μεταξύ των χωρών μελών και των νέων χωρών θα πρέπει να είναι βασισμένη στην αμοιβαιότητα. Πρέπει να ανοίξει το πρόγραμμα σε και σε άλλες χώρες, αλλά να συμμετάσχουν αυτές σε βάση αμοιβαιότητας. Σας ευχαριστώ κυρία μου, λέει ο πρόεδρος Μπούσεκ. Η κυρία Μίρκονεν. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να λάβω την ευκαιρία για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους θαυμάσιους ομιλητές και ιδίως στους Ιάπωνες προσκεκλημένους μας που ήλθαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξέφρασαν τις απόψεις των. Για μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία στην έρευνα και στη βιομηχανία μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Τώρα που έχουμε την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας σημαίνει ότι θα είναι ακόμα στενότερη η διασύνδεση και πολλές νέες ευκαιρίες θα έχουμε επίσης. Είμαι Φιλανδή η Φιλανδία είναι από τις χώρες εκείνες οι οποίες πάντοτε έχουν επενδύσει πολύ σε έρευνα και καινοτομία, βεβαίω όχι τόσο πολύ όσο η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι η Ιαπωνία πάντοτε επένδυσε πολύ σε έρευνα και ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία ε, επενδύει το 3,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της. Έχουμε βάλει και εμείς το στόχο στην Ευρώπη να φτάσουμε το 3. Όμως ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε καν το 2% του ΑΕΠ. Άρα μένουν πολλά πράγματα να κάνουν οι χώρες μέλη. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει όλες τις χώρες μέλη να πράξουν όπως η Ιαπωνία, να επενδύσει στην έρευνα και στην ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι αναγκαίο για το μέλλον μας. Είστε πραγματική ιστορία επιτυχίας. Πολύ ικανοποιημένες επίσης είμαστε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση του κοινού ερευνητικού προγράμματος ήταν 8 δισεκατομμύρια στο προηγούμενο ε, ΠΔΠ 80 μάλλον. Τώρα έχει προταθεί ε, να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια. Εμείς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή ζητούμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, να φτάσει στα 120 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η θέση μας. Θα τη διαπραγματευτούμε βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη. Αλλά επιθυμούμε να αυξηθεί η επένδυση, η δαπάνη στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Είμαι βεβαία ότι θα μας υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνεργασία μας με τρίτες χώρες όπως η Ιαπωνία στο μέλλον, διότι γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ποιότητα έρευνας και ανάπτυξης αυτή να έχει διεθνή χαρακτήρα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους ομιλητές που προσήλθαν σήμερα εδώ και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για όλες και όλους μας που εργαζόμαστε στον χώρο της έρευνας και ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Άλλος κανείς? Ε, εκ των μελών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε Μέντος, αξιότιμοι φιλοξενούμενοι μας. Σας ευχαριστώ για το χρόνο και την προσπάθεια για να παραστείτε στην Επιτροπή μας. Το προφανές μπροστά μας είναι η μελλοντική συνεργασία με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Εν γέννη αναφέρει σχετικά με αυτό ότι η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας είναι κρισίμου σημασία στα πλαίσια του ορίζοντα Ευρώπη. Εστιαστήκατε επίσης στον αντίκτυπο της συνέπειας και θέλετε προσέγγιση που βασίζεται στον αντίκτυπο και με συνεργασίες. Αναφέρθηκε η υπηρεσία σας σε εξοθολογισμό του προγράμματος. Οπότε διευκολύνονται οι άλλοι εταίροι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως να συμμετέχουν. μπορείτε να εξετάσετε διαφορετικές διεθνείς συνεργασίες. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Υποθέτω και κάτι άλλο. Αλλά φαντάζομαι δεν θα έχω απάντηση. Υποθέτω, λέγω, ότι πρόβλημα είναι πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός συγχρηματοδότησης. Θα πρέπει να περιμένω μέχρι τις 7 Ιουνίου για να ακούσω απάντηση. Ίσως όμως μπορείτε να μου πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία μου. Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δε, δε, λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας σήμερα. Έχουμε μακρύ ιστορικό συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ιαπωνίας. Είχαμε αρκετές αποστολές. Πήγαμε Πολλέ φορέ στην Ιαπωνία συμμετείχα σε μια τέτοια αποστολή, ήμουν τυχερή το 2013. Και χάρηκα που λαμβάνει η χώρα αυτή η συνεργασία. Χαίρομαι και όσον αφορά την αύξηση του προπολογισμού για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Στο Κοινοβούλιο προτείνουμε αύξηση. Δεν πήραμε αυτά που ζητήσαμε τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης πρότεινε κάποιο ποσό και ελπίζουμε τελικά φέτος να, να πάμε στο σωστό ποσό που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούστηκαν κάποιες ερωτήσεις, να προσθέσω κάποια στοιχεία που δεν θίγησαν ακόμα. Και εγώ έχω παρόμοια ερωτηματικά όπως αυτά που ετέθησαν από συναδέλφους μου ήδη. Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας που πράγματι έχει βελτιωθεί και έχει βελτιωθεί πολύ όσον αφορά την ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχει πραγματική συνεργασία βάσει συμπληρωματικότητα, συνεργασία μεταξύ χωρών, συνεργασία που βασίζεται επί αμοιβαιότητας και ε, μελλοντικής προπτικής. Ε, ερώτηση. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας στην οποία συμμετέχουμε, ότι θα εξακολουθούμε να προωθούμε την πολιτική χρήση της τεχνολογίας. Πώς είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία με τέτοιες χώρες θα είναι κάτι που βασίζεται επί του σεβασμού και θα χρησιμοποιείται βάση των ε, αξιών για, για, τις, ε, την ανθρώπινη, για των ανθρωπίνων αξιών που είναι κοινέ με την Ιαπωνία. Έχουμε ένα πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ανθρώπινα δικαιώματα και καμιά φορά συναργόμαστε με άλλε χώρε που δεν έχουν τι ίδιε αξίε όσον τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι σε αυτή τη συνεργασία θα λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστώ, κυρία μου, λέει ο πρόεδρο. Δεν ξέρω αν ζητάω στο λόγο από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Ο Επίτροπος σας απαντήσει στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Thank you very much, Chair, and thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ σας για τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω την κυρία Κεντρίκα. Θα είμαι λεπτομερέστερος σε μία-δύο εβδομάδες. Να σας διαβεβαιώσω για δύο πράγματα. Το πρώτο. Ποια είναι η δέσμευσή μου. Δεσμεύομαι να αυξήσω το ποσό που έχουμε σήμερα. Μέσω διεύρυνσης, μέσω συνεργασίας, μέσω συμμετοχής των χωρών. Να βελτιωθούν οι χώρες. Αυτή είναι προσωπική μου δέσμευση, την έχω επαναλάβει. Σύνθημά μας πρέπει να είναι η αριστεία. Αλλά να βοηθάμε και τους άλλους να φτάσουν στο επίπεδο της αριστείας, να γίνουν άριστοι. Αυτό το εστερνίζεστε, το ξέρω. Και είναι σημαντικότατο για το πρόγραμμα. Ελπίζω να έχω ευχάριστη έκπληξη όσον αφορά το πώς θα βοηθήσουμε όλους. Μετά μπορούμε να συζητήσουμε εκτενέστερα το θέμα. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τα πάντα τώρα, αλλά σας λέω ότι θα έχουμε σημαντική αύξηση, ουσιαστική αύξηση. Δεύτερον, η έκθεση Λαμή ετέθη στο ερώτημα. Από αναφέρονται χώρες όπως είναι ο Καναδάς και η Αυστραλία. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένες χώρες. Όμως, ήθελα να πω ότι η διεθνή συνεργασία πρέπει να είναι ανοιχτή και να είναι ανοιχτή όχι μόνο στα πλαίσια επιστημονικά και να, μην, να είναι διπλωματία επιστημονική, διπλωματία μέσω της επιστήμης. Έχουμε συνδεδεμένη χώρα την Τινησία. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα. Η Τινησία πολεμούσε για τη δημοκρατία. Έδωσε μεγάλη μάχη σε φρικτή ιστορική στιγμή και θέλαμε να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτό ήταν πολύ καλό. Το ίδιο κάναμε και με την Ουκρανία. Όμως θέλουμε και χώρες όπως ο Καναδάς να καλύπτεται. Ο Καναδάς που είναι μια υπέροχη επιστημονική χώρα. Μπορούμε να μάθουμε με ένα τους δε. Η απάντησή μου είναι ναι. Ο στόχος είναι κάτι που θα μου επιτρέψει να πλησιάσω χώρες όπως είναι ο Καναδάς, διότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Άρα χρειάζονται κριτήρια άλλα από αυτά που έχουμε σήμερα. Ούτω ώστε να μπορούμε να καλύψουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που δεν μπορώ να απαντήσω σήμερα είναι το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εξαρτάται το Ηνωμένο Βασίλειο από άλλες συζητήσεις, από διαπραγματεύσεις το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν εξαρτάται από μένα. Αυτό που εξαρτάται από εμάς, όχι από μένα, αλλά και από σας, είναι το εξής να έχουμε μια έννοια σύνδεσης που θα βοηθά άλλες χώρες να συμμετέχουν και να έρθουν μαζί μας. Αν στο μέλλον το Ηνωμένο και εμείς αποφασίσουμε για κάποια μελλοντική σχέση στις επιστήμες και ελπίζω ότι μετά από αυτή την αναταραχή να φτάσουμε σε ένα στάδιο που θα έχουμε μια μελλοντική σχέση και αν αυτό είναι εφικτό και αν διαπραγματεύσεις πάνε καλά και αν όλα πάνε καλά νομίζω ότι η θύρα είναι ανοιχτή. για το Ενωμένο Βασίλειο. Για πολλούς λόγους. Μας χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο και εμείς το χρειαζόμαστε. Θα είναι υποφελές και για τις δύο πλευρές. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό. Και θα σχεδιάσουμε όλα με μελλοντοστροφική μελλοντοστραφή προσέγγιση και θα προσπαθούμε να καλύψουμε και άλλες χώρες όπως ο Καναδάς. Είπατε και κάτι άλλο να εξετάσουμε τα, τους αριθμούς, πόσες άδειες ευρεσιτεχνίας ε, κλπ. Κυρία Καμπεζόν Ρούις. Σας ευχαριστώ που με συγχαρήκατε. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Σωστά τα είπατε. Όταν ήσασταν εισηγήτρια και ετοιμάζατε την έκθεσή σας, αυτή μας βοήθησε πολύ για τη στρατηγική μας, γιατί αφορούσε την ε, διεθνή συνεργασία. Αυτό υποστηρίζεται πάντα. Χρησιμοποίησατε μια λέξη πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης. Αμοιβαιότης είναι η λέξη. Δεν αφορά μόνο τις επιστήμες, αλλά πολλά από αυτά που κάνουμε. Χρειάζεται καλύτερη παγκοσμιοποίηση. Χρειάζεται περισσότερη αμοιβαιότητα. Και σήμερα οι σχέσεις μας δεν είναι πάντα αμοιβέ. Είναι ανοιχτή η Ευρώπη, αλλά καμία φορά άλλη δεν είναι ανοιχτή. Έχουμε περιπτώσεις όπου οι χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας, αλλά οι εταιρείε μας δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα δικά τους προγράμματα. Ή θα σας πω λοιπόν ότι πολιτικός πώς συμφωνώ μαζί σας. Η κυρία ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Όπως είπατε, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους, Πολύ δουλειά. Είναι πολύ καλό να ξέρει κάποιο ότι όλοι σε την αίθουσα και το Κοινοβούλιο παρέχουν υποστήριξη. Κυρία Βίρινγκ, αναφερθήκατε στη μελλοντική συνεργασία με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση για γνωστούς λόγους. Ελπίζω ότι θα έχουμε μελλοντική σχέση. Πάντα το έλεγα αυτό και αν σχεδιαστεί με έναν τρόπο που το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμμετέχει σαν τρίτη χώρα σε μια δίκαιη σχέση, θα είναι καλό. Θέλω να πω και το εξή. Όποια και θα είναι η πρόταση που θα υποβληθεί σε εσά, θα είναι δίκαιη. Όσον αφορά τη σχέση, τα ποσά, θέλω οι χώρες να συμμετέχουν και πρέπει να είμαι δίκαιο Δίκαιος και όσον αφορά το κόστος πόσο κοστίζει η οργάνωση του όλου θέματος, έχουμε διοικητικό κόστος, χρειάζεται μια δίκαιη σχέση, όπου να πληρώνουν το μεριδιό τους οι χώρες για τη σχέση. Πολύ γρήγορα. Για τη συγχρηματοδότηση, ο σχετικός μηχανισμός υφίσταται, είναι μια πραγματικότητα, έχουμε πολύ καλά παραδείγματα συγχρηματοδότησης, δεν έχω υπόψη μου κάποια σημαντική αλλαγή του μηχανισμού συγχρηματοδοτήσεως, θα σας δώσω λεπτομέρειες αργότερα. Κυρία Ματίας, θα μιλήσω πορτογαλικά. Ένα, δύο λεπτάκια πορτογαλικά. Κυρία Βουλευτή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου που παρίσταστε. Λοιπόν, αυτό που είπατε ήταν υπέροχο. Είπα την προηγούμενη φορά ε, ήταν για 100 εκατομμύρια και τελικά πέρασαν τα 80. Τώρα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 100 και το Κοινοβούλιο 120. Ελπίζουμε πάντα, ε, πάντα συζητάμε τα κονδύλια που πάνε στην έρευνα. Με ρωτήσατε αν στο μέλλον το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη θα έχει πολιτικούς σκοπούς. Ναι, πάντα αυτό ισχύει δεν υπάρχουν στατιωτικοί σκοποί του προγράμματος. Τίποτα λοιπόν δεν θα αλλάξει. Μου θέσετε και μια ερώτηση όσον αφορά τις αξίες. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτοί που συμμετέχουν, που συνεργάζονται μαζί μας, θα πρέπει να μοιράζονται μαζί μας τις ίδιες αξίες όπως και εμείς. Την αξία της ανθρώπινης ζωής, τη θεμελιώδη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βασικό όχι μόνο στον τομέα των επιστημών, αλλά σε όλους τους τομείς συνεργασίας. Διότι Εάν δεν γίνονται σεβαστές οι αξίες μας, τότε δεν είμαστε στο ύψο των περιστάσεων όσον αφορά τι εργασίε μα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε. Δεν χρειάζεστε καν διερμηνία. Μάλλον τα λέτε και πιο καλά στα πορτογαλικά από ό,τι στα αγγλικά, αν αυτό βεβαίω είναι δυνατόν. Αγαπητοί φίλοι, αυτό μου κάνει την ε, εξαιρετική πάσα από αυτή την εναρκτήρια σύνδο να περάσω στο επόμενο κομμάτι της συνεδρίασης. Έχουμε δύο πάνελ, δύο συνεδρίες. Θα ξεκινήσει να τα παρουσιάζει ο κύριος Σερουμπίκ που είναι πάρα πολύ ειδικό και κυρίως για τα θέματα της Επιτροπής ΤΟΑ είναι ε, σήμερα πρώτος αντιπρόεδρος, διετέλεσε όμως και κατά το παρελθόν πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ πρόεδρε. Είναι θαυμάσιο που μπορείτε να τα πείτε και στα γερμανικά. Ε, τώρα για τις μεταφράσεις μεταξύ Ιαπωνικών, Αγγλικών κλπ. πιο εύκολα είναι. Χαίρομαι διότι η επαφή με το φόρουμ STS είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρόκειται για το Παγκόσμιο Φόρουμ Οικονομικών και ε, εκεί το φόρουμ αυτό που εντάσσεται είναι πολύ σημαντικό για την τεχνολογία και πολύ σημαντική συνεργασία μαζί του. Γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στους πολίτες μας και βέβαια τα 100 δισεκατομμύρια για τα οποία μιλούμε τώρα δεν αρκούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και τον γεωργικό τομέα, διότι και ο γεωργικός τομέας χρειάζεται νέους στόχους, νέες δραστηριότητες και τεχνολογίες. Θα προτείνω να στοχεύσουμε ιδίως στον δεύτερο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης, ασφάλεια τροφίμων, τον 6 ε, υγιεινή, καθαρό νερό και των επτά που είναι ανανεώσιμες ενέργειες που είναι και στην καρδιά των ενδιαφερόντων της Επιτροπής μας. Θα είναι εύκολο να συζητήσουμε και με τους ανθρώπους ε, το, της Επιτροπής Γεωργίας ότι πρέπει να κάτι να κάνουμε για τους νέους γεωργούς και πρέπει κάτι να κάνουμε και στον τομέα της ανάπτυξης ιδίω υπέρ της Αφρικής όπου πρέπει να εξασφαλίσουμε οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, με τη δουλειά τους δηλαδή, και να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Τώρα μιλούμε πλέον για αυτοκίνητα που οδηγούνται μόνα τους. Όμως πολύ πιο σημαντικό και ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε τις υποδομές μεταξύ αυτών την ε, τεχνητή νοημοσύνη και να τα εγκαταστήσουμε, να τα εντάξουμε όλα αυτά στις τεχνολογίες μας. Σημαντικό αυτό για να φτάσουμε μέχρι και τις περιφέρειές μας, ώστε οι τεχνολογίες αυτές να μπουν παντού, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Ξέρω ότι έχουμε τώρα την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία μπορεί να προσφέρει πολλά προϊόντα και υπηρεσίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει πολλά στην Ιαπωνία. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε χέρι με χέρι ε, σε μια σημαντική ανάπτυξη. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων και στο STS Forum και στη ΣΤΟΑ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε που μας επιτρέπεται να προχωρήσουμε με συνεπή τρόπο στην κατεύθυνση αυτή. Πάρτε τα social media στα οποία συμμετέχετε και πέστε στον κόσμο ότι επιστήμη και τεχνολογία πρέπει να μπουν στις πρώτες πρώτες προτεραιότητες της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίω. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και εγώ λέει ο πρόεδρος ε, Μπούσεκ Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές για την αναρκτήρια συνεδρία. Τώρα σας παρακαλώ να δεχτείτε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, στη διάρκεια του οποίου θα προσκαλέσω τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο πρώτο πάνελ, που είναι η κυρία Ρουσό, ο κύριος Μακκίναλ, ο κύριος Τουμπάτσι και ο κύριος Ιρίνο και ο καθηγητής Μπουργκινιόν που θα είναι ο διευθυντής της συζητήσεως και είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου Ερευνών. Αρχίζουμε, λοιπόν, μάλλον αλλάζουμε θέση στο, εδώ στο έδρανο του Προεδρείου και αμέσως μετά θα αρχίσουμε. Ladies Κυρίες και κύριοι, έχω αναλάβει το καθήκον να, παρουσιάσω την πρώτη συνεδρία με τίτλο «Μίζωνες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, συνεργασία στο πλαίσιο του ορίζοντα Ευρώπη, μια Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο μέσω του φόρουμ STS». Έχουμε μια ομάδα μιλητών που θα απευθυνθούν στο κοινό για το θέμα αυτό. Πρώτη η κυρία Κριστίνα Ρούσο Η κυρία Χριστίνα Ρούσο εργάζεται στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή είναι Διευθύντρια Διεθνού Συνεργασία από τον Ιούλιο του 2013. Αρμόδια για την πρόθεση της έρευνας καινοτομία και τη σχετική συνεργασία ε, με τους Διεθνεί εταίρους για την ενίσχυση της επιστημονική αριστείας και τη ελκυστικότητα τη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, καθηγητά Μπουργκίνιο και καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι δύσκολο ε, να πάρει κανείς το λόγο μετά από μια τέτοια πλειάδα ε, ομιλητών. Ακούσαμε τον κύριο Μοέδας και άλλους σημαντικούς ομιλητές. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ε, επειδή πιέζει ο χρόνος, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω, θα είμαι σύντομη και θα πω μόνο λίγα πράγματα εν αγωγής για τη συνεδρία αυτή που έχει τον τίτλο «Μίζωνες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, η συνεργασία μέσω του Ορίζοντα Ευρώπη, η Ανοιχτή Ευρώπη στον κόσμο, μέσω του Φόρουμ STS». Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι το, το ένατο ε, πρόγραμμα πλαίσιο, Ορίζοντα ε, Ευρώπη λέγεται πλέον, αυτή είναι η πρόταση, το είπατε, και προηγουμένως ε, έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις, μακές, τις ε, βασικές κοινωνικές αλλαγές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Έχουμε εργαστεί σκληρά για να προετοιμάσουμε αυτό το σχέδιο Horizon Ευρώπη. Είχαμε διαβουλεύσεις με τους ε, ενδιαφερομένους φορείς, με την επιστημονική κοινότητα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης προσεγγίσαμε τους πολίτες αλλά και τους επιστήμονες για να κατανοήσουμε πού έγκυνται αυτές οι μείζονες προκλήσεις που θέλουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε για να προωθήσουμε το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη για την καινοτομία και την επιστήμη. Ευρεία η διαβούλευση. Όπως γνωρίζετε, μπορώ να σας δώσω και λεπτομέρειες, 7 Ιουνίου θα εγκριθεί το Ορίζον Ευρώπη, αλλά τη στιγμή της έγκρισης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου έγινε μια παρουσίασή του, οπότε μπορώ να σας πω δύο πράγματα. Θα έχει τρεις πυλώνες το πρόγραμμα. Ο πρώτος πυλώνας, και σε αυτόν θα εστιάσω, παγκόσμιες προκλήσεις. Και οι άλλοι δύο είναι ανοιχτή επιστήμη και ανοιχτή καινοτομία. Παγκόσμιες προκλήσεις. Ο πυλώνας αυτός έχει σχεδιαστεί ιδιαίτερα και συγκεκριμένα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που κινούμε τους επιστήμονες, τους πολίτες. Είναι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και πρέπει ε, να ε, προωθήσουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, καλύπτοντα τομεί, ε, την υγεία, την ασφάλεια τροφίμων, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, το κλίμα, την ενέργεια κινητικότητα, χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα, οικολογική κοινωνία και σημαντικέ άλλε δραστηριότητε για του τομεί που οποίου στηρίζεται η οικονομία μα και η κοινωνία μα. Αυτό που θεωρούμε σημαντικό είναι αυτά να γίνουν από κοινού, στο πλαίσιο επιστημονική συνεργασία. Σα είπα θα είμαι σύντομη. Βέβαια, θέλω να πω δύο λόγια για τη στρατηγική συνεργασία μα με την Ιαπωνία. Εφόσον βρισκόμαστε εδώ στο πλαίσιο μια συζήτηση με το Φόρμες STS. Η Ιαπωνία για εμάς, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας επιστημονικός εταίρος για τη συνεργασία μας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Αντιμετωπίζουμε με την Ιαπωνία τις ίδιες προκλήσεις. Γύρανση του πληθυσμού, ενεργειακή ασφάλεια, πρόσβαση σε σημαντικές πρωτεσίλες, αύξηση της ευμερίας των πολιτών. Έχουμε επίσης παρόμοια προσέγγιση σε ό,τι αφορά βασικούς διεθνείς στόχους. Έχουμε λοιπόν τακτικούς διαλόγους πολιτικής μεταξύ Απωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τη μεικτή ε, διευθύνουσα επιτροπή η οποία ε, συνεδρίασε πρόσφατα. Έχουμε ε, ενδιαφέροντα για το κλίμα, την ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, κλιματική έρευνα, αυτοματοποιημένη οδήγηση κτλ. Είναι σημαντική τομή όλοι αυτοί. Από κοινού με τους επιστήμονες και της Απωνίας αλλά και άλλων χωρών του κόσμου συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αυτές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. So the Επόμενος ομιλητής. Ο κ. Γιάσου Κάτσου τελεξιστικός αντιπρόεδρος της ΤΕΤΡΟ η οργάνωση εξωτερικό εμπόριο της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο 2017 ήταν υποδιευθυντή γενικός για εμπορική πολιτική στο, στο Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας του ΜΕΤΗ. Έχει ε, πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Τόκιο και ήταν εμπορικό σύμβουλο στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Πρεσβεία τη Ιαπωνία και ήταν επικεφαλής του γραφείου Σιγκαπούρη, υπεύθυνο για Οκεανία και Ασία και εκπροσωπούσε το ΜΕΤΙ εκεί. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Γεια σας, είναι το όνομά μου. Αντιπρόεδρος του Τζέτρο. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσω. Η Τζέτρο, λοιπόν, ο Οργανισμός Εξωτερικού Μπορείου της Ιαπωνίας, είναι οργάνωση της κυβερνήσεως της Ιαπωνίας και προωθεί αμφίδρομο εμπόριο και επενδύσεις μεταξύ Ιαπωνίας και υπολείπου κόσμου. Έχουμε παγκόσμιο δίκτυο που καλύπτει 74 περιφερειακά γραφεία σε 54 χώρες. Μεταξύ αυτών 14 γραφεία έχουμε σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Το προσωπικό της Τζέτρο Βρυξελών συμμετέχει επίσης στο σημερινό φόρουμ Ευρύνεται το δίκτυο και συμβάλλουμε στις εμπορικές δραστηριότητες του ε, φόρουμ STS στον κόσμο. Η, η οργάνωση προθήσεως εμπορίου και επενδύσεων ελπίζει ότι η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσουν την καινοτομία στο μέλλον και θα βελτιωθεί η σχέση και έτσι οι δύο περιφέρειες θα διευκολύνουν το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ τους, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπροσωπώ την οργάνωση εμπορίου ε, της Ιαπωνίας και της καινοτομίας και θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας από την έποψη των παγκοσμίων προκλήσεων. Το πρώτο θα πω, η συμμετοχή του Τζέτρο στο διεθνές εμπόριο και στην, εκ, και στην καινοτομία. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την τέταρτη ε, επανάσταση. Υποστηρίζουμε πρόγραμμα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα αν αυτά τα θέματα ε, καθοδηγήσουν τι μελλοντικέ συζητήσεις. Οι παρόσε βιομηχανικές δομές αλλάζουν με δραματικό τρόπο λόγω της τέταρτη βιομηχανικής επανάστασης και η τάση δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς να λάβουμε υπόψη τι καινοτομίε. Η τέταρτη αυτή η επανάσταση δημιούργησε νέου τομεί επιχειρηματικότητα. όπως είναι το διαδίκτυο, ε, η οικονομία στο διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη και, τα, και η ρομποτική. Όλα αυτά θα αλλάξουν το παραδοσιακό επιχειρηματικό πλαίσιο. Και σαν οργάνωση και εμείς θα πρέπει να συμμορφωθούμε και να προσαρμοστούμε στην τάση. Και γι' αυτό κάναμε προσπάθεια η οργανώσεως μιας έκθεσης με αυτά τα θέματα και βοηθούσαμε τις νεφείς επιχειρήσεις σχετικά με την καινοτομία και να διαδοθεί η επιχειρηματικότητα ιαπωνική ε, υπεράκτια. Οι νεοφυείς εταιρείε δημιουργούν νέα προϊόντα και υπηρεσίε και προωθούν την καινοτομία στην κοινότητα, στην κοινωνία. Και θέλουμε αυτό να γίνεται σύντομα και να διατίθεται τα προϊόντα και στην εγχώρια αγορά αλλά και στη διεθνή αγορά. Αυτό είναι ο στόχος. Όσον αφορά του τομεί δραστηριοτήτων, όπως προανέφερα, συμμετέχουμε στη Διεθνή Έκθεση για Αυτοματισμό τεχνολογία πληροφορικής και τηλεπικοινωνίες, το SEBIT, στο Ανόβερο, στη Γερμανία. Ε, το Μάρτιο του 2017 συμμετείχαμε. Η Τζέτρο παρουσίασε εκθέματα την Ιαπωνία, συμμετέχοντας στη SEBIT. Η πρόοδος βασίζεται στη νέα τεχνολογία, όπως ε, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή τεχνολογία. Τα θέματα τα ενεργειακά και η προκλήση του περιβάλλοντο μπορούμε τη νέα τεχνολογία να αντιμετωπιστούν και η γύρανση του πληθυσμού. Πώ την καινοτομία να την ταιριάξουμε, να προωθήσουμε τη νέα τεχνολογία. Η Τζέτρο θα εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε συνεργασία καινούρια, να δημιουργεί νέε προπτικές, νέα τεχνολογία επιλύοντας κοινωνικά προβλήματα. Η Τζέτρο είχε δραστηριοποιηθεί σχετικά με την καινοτομία, αυτό που συζητάμε σήμερα. Θα πρέπει να πέσουν οι φραγμοί μεταξύ εργαστηρίου και εταιρεία. Όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείε, αλλά και τι νοφεί επιχειρήσει, Οπότε να αλλάξει το οικοσύστημα τη καινοτομία, να υπάρξει καλύτερη επαφή μεταξύ εργαστηρίου και επιχειρήσεις. Για την καινοτομία, να πω ένα παράδειγμα. Το πρόγραμμα και το Τζέτρο είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει, όπου οι νεφείς γιαπωνικές επιχειρήσεις μπορούν να εργαστούν στο εξωτερικό και πρώτα λαμβάνουν κατάρτιση και μαθαίνουν για επιχειρηματικά μοντέλα στην Ιαπωνία και μετά πάνε ε, σε όλο τον κόσμο σε άλλες χώρες. Πάνε στο Σεντζέν στην Κίνα, στη ΣΥΠΑ κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία θα αναπτυχθούν μέσω της καινοτομίας αυξάνουν τις επενδύσεις και το εμπόριο. Η Τζέτρο έχει στόχο την Ευρώπη για πρώτη φορά και θα χρησιμοποιήσει τις νεφοείς επιχειρήσεις που θα αποσταλούν στην Ευρώπη το φθινόπωρο. Και η Ιαπωνική κυβέρνηση βοηθάει τις νεφοείς επιχειρήσεις. Εφαρμόζοντας κυβερνητικές, κυβερνητικές πολιτικές με διάφορες εκδηλώσεις. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια εκδήλωση η JetRo θα έχει το περίπτωρο της Ιαπωνίας στην έκθεση. Σε τέσσερα χρόνια είχαμε συμμετάξει στο συνέδριο για την κινητή τεχνολογία. Στον τομέα της κινη... κινητής τεχνολογίας. Αλλά θα γίνει στην Ισπανία τον επόμενο Φεβρουάριο μια τέτοια εκδήλωση. Θέλουμε εκδηλώσεις για να προωθούμε την καινοτομία. Επαφές μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών και νοφιών επιχειρήσεων. Θα παίξει ρόλο η καινοτομία για να λύσει προβλήματα και να διερευνά νέους τομείς στην τεχνολογία και στη βιομηχανία. Γίνονται όλο και σημαντικές οι νεοφυείς εταιρείε και στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη. Πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερε προσπάθειες για να δημιουργήσουμε ευκαιρίε επιχειρηματικέ για τέτοιε εταιρείε. Θα ήθελα Κλείνοντα να σταματήσω αναφερόμενο σε νέα δραστηριότητα και πρόγραμμα υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Στην ΖΕΤΡΟ ελπίζουμε να συνεχιστεί η συνεισφορά μα στον τομέα επιστήμης τεχνολογία μέσω του φόρουμ STS. δρόκα σαν γέφυρα που συνδέει τη παγκόσμια επιχειρηματικότητα, τα πανεπιστήμια και του διαμορφώντε στην πολιτική. Ελπίζω ότι το σημερινό εργαστήριο θα αποτελέσει καταλήτη για περαιτέρω ενίσχυση τη συνεργασία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Ο πρόεδρος Μπουργκινιό, σας ευχαριστώ κύριε Ήρινο. Ακολουθεί ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τσουμπάτσι, πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Προηγμένης Τεχνολογίας. Με παρακάλεσαν να είμαι πολύ σύντομο στις παρουσιάσεις που κάνω τον. Ε, προσωπικότητων. Δεν θα υπενθυμίσω όλες ε, τις ε, δραστηριο, προηγούμενες δραστηριότητες και τίτλους σας μεταξύ αυτών και την εταιρεία Sony. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγική σας παρατήρηση. Θα ήθελα σήμερα να σας εξηγήσω την ε, κατάσταση στην Ιαπωνία και τις δραστηριότητες για την έρευνα και την ενέργεια. Μετά από την βιομηχανική επανάσταση, η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν αναπτύξει την οικονομία με μαζική χρήση φυσικών πόρων και κεφαλαίων. Από την άλλη μεριά, αυτά έχουν προκαλέσει και σοβαρά ζητήματα, όπως καταστροφή του περιβάλλοντος και ε, η κατάχρηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή είναι επίσης ένα ζήτημα που επιζητεί την επίλυσή του. Έχουν γίνει διεθνείς προσπάθειες για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στη βάση του πρωτοκόλλου του Κιώτο η Ιαπωνική κυβέρνηση έχει σχεδιάσει την σχετική πολιτική της βάζοντας προτεραιότητες στα εξής. Ασφάλεια ενεργείας, οικονομία και, και ε, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια περιβάλλον. Στη Συμφωνία των Παρισιών αποφασίστηκε το 6% να μειωθεί κατά το 6% μέχρι το, 20, το 2030. Για να γίνει αυτό χρειάζεται αυξημένη προσφυγή σε ανανεώσιμες ενέργειες. Ωστόσο στην Ιαπωνία βρισκόμαστε ακόμα στο 15% της συνολικής παραγωγής ε, ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες ενέργειες. Η κυβέρνησή μας προ λίγων ημερών ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2030 σκοπεύει να φτάσει την αναλογή αυτή στο 24% και να γίνουν και κυρίαρχη πηγή ενέργειας στο μέλλον. Ωστόσο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά ε, εμπόδια. Το αρχικό επενδυτικό κόστος είναι υψηλό. Ε, προβλήματα υπάρχουν και με την διασυνδεσιμότητά τους με τα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς τη ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν και συγκεκριμένα εμπόδια στην ίδια την Ιαπωνία. Είμαστε νησιωτική χώρα. Η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματο από γειτονικέ χώρε οικονομικά είναι ανέφικτη. Πολλές φυσικές καταστροφές προκαλούν σημαντικά ζητήματα ε, ασφάλειας στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά. Οι προκλήσεις αυτές δεν μπορούν να λυθούν από μια μονάχα, μονάχα εταιρεία ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεργαστούν σε μεγάλη κλίμακα. Όπως είπε προηγουμένως ο κύριος ε, Σατός στην προηγούμενη ε, συνεδρία, κάνουμε σημαντική προσπάθεια για να αναπτύξουμε τις σχετικές τεχνολογίες. Κάνουμε έρευνα και ανάπτυξη για την ενέργεια εδώ και πολλά χρόνια. Μετά από τον πρόσφατο σεισμό το 2011 και την πυρηνική καταστροφή δημιουργήσαμε το Ινστιτούτο το, στη Φουκουσίμα για την πυρηνική ενέργεια. Εδώ αυτό ασχολείται με την αντιμετώπιση τριών προκλήσεων. Δημιουργία ενέργειας, αποθήκευση και μεταφορά και εξοικονόμηση ενέργειας. Για τη δημιουργία της ενέργειας διεξάγουμε έρευνα με φωτοβολταϊκά τόξα για την παραγωγή ενέργειας. Για παράδειγμα, αναπτύσσουμε κύτταρα ε, φωτοβολταϊκά με αποδοτικότητα 30%. Προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε επίσης την παραγωγή ενέργειας με αισθητήρε που προβλέπουν ε, την ηλιοφάνεια και την συγκατεύθυνση των ανέμων. Το ίδιο κάνουμε και με κύτταρα υδρογόνου. Ιδίως για το υδρογόνο χρησιμοποιούμε και, άλλες, και άλλους χημικούς τύπους και, και υλικά όπως αμμονία που έχουν και ε, πλονεκτήματα και μειονεκτήματα. Διερευνούμε τους καλύτερους τρόπους χρήσης για κάθε έναν από τους φορείς αυτούς παραγωγής ενέργειας. Συνεργαζόμαστε άλλωστε και με μεγάλες εταιρείες στην Ιαπωνία για να φτιάξουμε συστήματα μεταφοράς των ε, ανανεώσιμων ενεργειών. Για να εφτάσουμε σε μια βέλτιστη παραγωγή ενέργειας και θέρμανση. Χρειάζεται επίσης και η συλλογή και αποθήκευση της ενέργειας μέσω των υφισταμένων δικτύων. Παράγουμε επίσης ημιαγωγούς με silicon carbide και στις, στη βάση των τεχνολογιών αυτών. Ελπίζουμε να γίνουμε πραγματικά πόλος για τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες, στέλνοντας ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για το πρόγραμμα Horizon της Ευρώπης και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε κάνουμε άλλο, εξάγουμε άλλωστε και κοινέ έρευνες με το Ινστιτούτο Fraunhofer, με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το Κέντρο Ερευνών των Κάτω Χωρών και ούτε καθεξής. Και επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με όλους αυτούς τους φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for very interesting πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε στον τελευταίο μιλητή για τη δεύτερη αυτή συνεδρία, τον κύριο Χέντρι Μακίνελ, πρόεδρο της Moody's Corporation. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα. Εγώ αισθάνομαι πιο καλά στο να συμμετέχω σε ε, συνεδρίες ερωταπαντήσεων. Ε, δεν προτιμώ να ε, εκφωνώ ομιλίες, αλλά τέλος πάντων. Μια ερώτηση ίσως θα μπορούσε να είναι τι ξέρει για την παγκόσμια υγεία και περίθαλψη ο πρόεδρος της Moody's Corporation. Για να απαντήσω πρέπει να σας πω ότι πήρα διδακτορικό στην ηλικία των 24 ετών από το Στάνφορντ. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο να μπει κανείς τότε. Το Στάνφορντ πήγε στη ΒΕ, ε, στην πολυμορφία και τότε ήμουν ε, ε, μπορούσα να πάω και στο Στάνφορντ και στο Χάρβαρντ και επέλεξα το Στάνφορντ τέλος πάντων στα 24 αποφάσισα να προχωρήσω με μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Αλλά πρώτα να αποκτήσω μια εμπειρία εργασιακή. Πήγα στη Pfizer λοιπόν, στην Ιαπωνία. Δύο χρόνια έμεινα εκεί. 36 χρόνια μετά Ήμουν διευθύνων σύμβουλος και παρετήθηκα. Ήμασταν μια εταιρεία φαρμακευτική με τη μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα και έχω μάθει πολλά πιστεύω ήδη. Πρέπει να σας πω επίσης ότι δεν είμαι μόνο ε, ε, ειδικό για αυτά τα θέματα λόγω της επαγγελματική μου ε, δραστηριότητας αλλά και για το ότι έχω δει τα διαφορετικά υγειονομικά συστήματα, συστήματα υγεία τεσσάρων βασικών χωρών και έχω σκεφτεί πολύ το θέμα χωρίς όμως να μπορώ να πω κάτι καλύτερο από αυτό που είπε ο Μαχάτ Κάντι όταν η πρώτη φορά ήρθε στο Λονδίνο. Ο Βρετανικό τύπο είχε ενθουσιαστεί με, το μοναδικό αυτό, τη μοναδική αυτή προσωπικότητα που ήταν δεσμευμένο να προχωρήσει σε μη βίαιε μεταρρυθμίσει ε, στην Ινδία. Βγαίνοντα μια μέρα από το αυτοκίνητο, υπήρχαν κάποιοι φωτογράφοι, ρεπόρτερ, κοντάκι και κάποιο ε, του φώναξε μια ερώτηση και η ερώτηση ήταν τι άποψη έχετε για το δυτικό πολιτισμό και ο Μαχάτμα σκέφτηκε για ένα-δυο λεπτά και είπε νομίζω θα ήταν καλή ιδέα. Άρα η εμπειρία μου με τέτοιου είδου ερωτήσει, τι πιστεύω για, όπω να πιστεύω για τα συστηματικές θα έλεγα ναι, καλή ιδέα θα ήταν, διότι δεν ξέρω κάποια χώρα που να είναι ικανοποιημένη με το σύστημα δημόσιας υγείας που έχει, ακόμη και αν υπάρχουν βέβαια διαφορετικά μοντέλα ανά τον κόσμο. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια ε, η οποία έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και δεύτερον, τιμή ε, τότε οικονομική της υγειονομικής περίθαλψης. Ε, υπάρχουν προβλήματα με την πρόσβαση που είναι πολύ εμφανή. Τα έχω δει και εδώ και στην Ποσαχάρη Αφρική και έχω ταξιδέψει πολύ Έχω υπηρετήσει και ως σύμβουλος ε, του George W. Bush ε, για τα θέματα υγείας ε, και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι αυτοί που χρειάζονται πρόσβαση στην υγειονομική πέθαλψη πρέπει να την έχουν και πρέπει να τα αποκριθούμε και στις μεταδοτικές νόσους, στη μεγάλη αυτή μάστιγα για την Αφρική. Ξέρω επίσης ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα η υγειονομική περίθαλψη με την επιστηστική βοήθεια. Δεν μεταφέρεις ε, τρόφιμα σε κομβόι και τα δίνεις στον κόσμο. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, θέλουν να φροντίσουν αυτούς που ε, πάσχουν από αυτά τα μεταδοτικά νοσήματα, φυματίωση, ελονοσία, HIV, AIDS κτλ. Εμείς δημιουργήσαμε ένα Ινστιτούτο για τα μεταδοτικά νοσήματα ε, το οποίο εδράσει στο Πανεπιστήμιο Μακάρ, γιατί θεώρησαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τοπική προσπάθεια ε, και η κοινωνία να συμμετέχει με στόχο να εκπαιδεύσουμε εκατοντάδες που αυτοί θα εκπαίδευαν χιλιάδε χιλιάδες και οι οποίοι θα ε, φρόντιζαν εκατομμύρια. Δέκα χρόνια ε, το κάνουμε ήδη 2000 ε, Έχουμε, είναι μη κερδοσκοπικό ε, ίδρυμα αυτό και τώρα εκπαιδεύουμε 25.000 επαγγελματίε του κλάδου της υγείας από 27 διαφορετικές χώρες και Αυστραλία και και υπάρχουν χιλιάδες ε, που ε, πλέον θεραπεύουν εκατομμύρια και στην Αφρική κυρίως βέβαια. Ε, το βασικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι ναι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας και της προστότητας. Αφού καταλάβουμε τι έγινε πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ έχω κάποιες δυνατότητες και έχω κάνει διάφορα πράγματα. Αν πάει κάποιος σε αυτό το Ινστιτούτο Μεταδοτικών ε, Νοσημάτων θα επισκεφθείτε το MKC που με μεγάλη περηφάνεια θα σας το δείξει ο κόσμος ε, για την ε, μέρημνα των ασθενών και την το McKinnell Knowledge Center, Knowledge Center, δηλαδή αντί να είμαι άνθρωπος πλέον έχω γίνει κτίριο. Σας ευχαριστούμε. Πολύ καλή αυτή η σύστασή σας προς δράση. Ήταν ευπρόσδεκτη. Μπορούμε να ακούσουμε λίγες ερωτήσεις. Έχουμε μείνει πίσω χρονικά και ξέρετε ότι εδώ βρισκόμαστε σε ευρωιαπωνική περιπέτεια και είναι προϋπόθεση και προαπαιτούμενο να είναι στην ώρα της Ιαπωνέζης. Να τελειώσουμε στην ώρα μας. Ερώτηση από το κρατήριο υπάρχει. Ουδεμία ερώτησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές για τη συνεισφορά τους και θα έχουμε την νέα ομάδα ομιλητών τώρα για το επόμενο τμήμα της συνεδριάσεως. Υποτίθεται ότι θα προείδρευα. Θα προεδρεύσω και του τρίτου τμήματος. Ας έρθουν η κυρία Μόλτσιτς, Σέρα Γκέλντιν, Τζούντι Μάξτον και Μότο Κοκότον. while the speakers are coming, since I'm really under pressure of time, so let's... Κοιτάξτε, έχουμε πίεση χρονική ε, να πω κάποια πράγματα εν είδη εισαγωγή αυτού του τμήματος συνεδριάσεως. Λοιπόν, δεν θα με ακρηγορήσω. Ο τίτλο είναι έρευνα με βάση την περιέργεια. Πώ ορίζον Ευρώπη μπορεί να συμβάλλει σε νέες ανακαλύψεις επιστημονικές. Εντάχει να πω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η έρευνα είναι πραγματικά ένα οικοσύστημα το οποίο εδράζεται επί της υποστηρίξεως που πρέπει ποικιλοτρόπως να διατίθεται. Ένας τρόπος είναι ο τυπικός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας να, να προσλαμβάνει συμβασιούχους για συγκεκριμένα προγράμματα. Υπάρχει και άλλος τρόπος υποστήριξης έρευνας ε, μέσω δικτύων και τα δίκτυα είναι σημαντικότατα για τη διεθνή συνεργασία διότι πράγματι ε, εντοπίζονται έτσι συγκεκριμένοι στόχοι, ερευνητικοί, κοινοί στόχοι. Μετά υπάρχει και η επαναλαμβανόμενη υποστήριξη που είναι πολύ σημαντική, ουσιώδη για τα εργαστήρια. Και τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό, διότι έχουμε ανθρώπου που κάνουν την έρευνα. Δεν είναι μόνο οι θεσμοί που κάνουν την έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμο να έχει κάποιο είδου θέση, εργασία σε διάφορα ε, επίπεδα καριέρα, σταδιοδρομία. Να έχουμε πάντα υπόψη λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το ερευνητικό οικοσύστημα. Δεύτερο σημείο που θέλω να πω. Λοιπόν, η έρευνα με βάση την καριέρα συνδέεται με ερευνητικά προγράμματα και προτάσεις που μπορεί να υποβάλει κάποιος σε διάφορους φορείς. Πρέπει να δεχτούμε και κάτι άλλο. Το έθεσε το παράδειγμα η Ιαπωνία με το GST, την υπηρεσία για επιστήμες και τεχνολογία που έχει η Ιαπωνία αλλά ακόμα και αν εντοπίσεις κάποια γενικά προβλήματα και πάλι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτωθεν προσέγγιση για να απαντήσεις τα προβλήματα και να βασίζεται επί της πρωτοβουλίας των ερευνητών αφού ερευνήσεις ε, ποιε είναι οι προτεραιότητες. Τέλος, εξίσου σημαντικό και αυτό, ε, πώς μπορείς να διασυνδέσεις την έρευνα με βάση την περιέργεια με αποτελέσματα και αντίκτυπο ο Επίτροπος Μέντες είπε ότι αντίκτυπος είναι για το ορίζον Ευρώπη βασική λέξη. Ακόμα κι αν ο αντίκτυπος δεν είναι κριτήριο την επιλογή προγραμμάτων και πάλι πρέπει να θέλουμε να έχουμε αντίκτυπο και αποτελέσματα και να συνοδεύουμε σωστά τους ερευνητές για να βελτιστοποιούν τα αποτέλεσμα του αντίκτυπου. Μπορεί να το κάνουν αυτό βάσει δικών τους πρωτοβουλειών αλλά με άλλο τρόπο. Το θέμα της διασύνδεσης έρευνας και με καινοτομία ακριβώς και ο τρόπος αντιμετωπίζεται με βάση τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα. Αυτά ήθελα να πω είναι είδη Η Βανέσα Σμόλτσιτς έχει το λόγο. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα ε, είναι στο τμήμα ερευνών του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ στην ε, Κροατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω το πρόγραμμά μου εδώ. Ετοίμασα, όπως βλέπετε, και κάνα δύο διαφάνειες οι οποίες θα συνοδεύσουν την ομιλία μου. Ε, έχω χορηγία, υποτροφία του ERC που σχετίζεται με ένα πρόγραμμα και αφορά την αστροφυσική και κάνω την έρευνά μου στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ. Να τονίσω ότι ήταν από τα προγράμματα, τα πρώτα προγράμματα ΕΡΣΥ που ανετέθη στην Κροατία και έχουμε πέντε τέτοια προγράμματα στην Κροατία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω παρουσιάζοντας τον εαυτό μου κάπως καλύτερα. Θα το κάνω αυτό στα πλαίσια της διαφάνειας, ανοιχτής προσέγγισης που αναφέρει και σήμερα. Η σταδιοδρομία μου ήταν πολύ διεθνή στο πανεπιστήμιο, στον πανεπιστημιακό χώρο και αυτό απαιτεί για να έχει κανείς μια σταδιοδρομία επιτυχή στο πανεπιστήμιο, διότι η μετάδοση της γνώσης σε διεθνές περιβάλλον μεγιστοποιείται, σε ένα ανοιχτό περιβάλλον μεγιστοποιείται. Το Masters, το οποίο στην Κροατία, στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεπ, όπου και εκεί εργάζομαι, σαν ε, καθηγήτρια και μετά πήρα το διδακτορικό μου στο Ινστιτούτο Max, ένα από τα Ινστιτούτα Max Planck στη Γερμανία. Μετά από αυτά είχα διάφορες, ε, είχα διάφορες θέσεις στο Caltech, στις ΗΠΑ ε, και στην Ευρώπη επισκέπτε καθηγήτρια και στην Αυστραλία. Οπότε ταξίδευσα εκτενώς και το 2013 μετά περίπου από 10 χρόνια σταδιοδρομίας εκτός Κροατίας επέστρεψα εις Κροατία. Η έρευνά μου ερευνά ένα τομέα Τη αστροφυσικής, τη παρατήρηση, Τι σημαίνει αυτό. Χρησιμοποιούμε τα τηλεσκόπια, τα καλύτερα τηλεσκόπια στον κόσμο. Γιατί, για να παρατηρούμε τμήματα του γαλαξία του ουρανού και η τεχνολογία είναι τόσο προθυμένη τώρα που συλλέγουμε πάρα πολλά στοιχεία πρέπει να εξεργαστούμε. Άρα είναι επιστήμη του big data. Πάρα πολλά στοιχεία. Παρατηρούμε τον ουρανό με τα καλύτερα τηλεσκόπια στον κόσμο. Αυτού του είδου η έρευνα απαιτεί πολλή έρευνα σε διεθνή ε, σε διεθνές επίπεδο και μεγάλες ομάδες που ξεχάζονται τα στοιχεία. Στις ομάδες που εργάζομαι έχουμε περίπου 100-200 ανθρώπους ανά ομάδα και τα μέλη της ομάδας είναι από όλο τον κόσμο. Ε, πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό του ERC, του οποίου ηγούμε, σχετίζεται με τη μελέτη διαφόρων πτυχών της εξελίξεως των γαλαξιών είναι παρατηρητική κοσμολογία. Είναι πολύ ενδιαφέρον τομέας. Στόχος, να μελετήσουμε κάποιες πτυχές του πώς αναπτύσσονται οι γαλαξίες σε κοσμικό χρόνο από τη γέννηση του σύμπαντος μέχρι σήμερα. Είναι επίκαιρο το πρόγραμμα και είναι σημαντικό αυτό διότι έχουμε προθυμένη τεχνολογία όσον αφορά τα εργαλεία σε όλο τον κόσμο, τι τελευταίε δεκαετίε σε όλο τον κόσμο. Σημαντικές εξέλιξει τεχνολογικέ. Όταν πήρα τη χορηγία του ERC, ε, μας επέτρεπαν τα μέσα, τα τεχνικά, να κάνουμε άλματα προόδου επιστημονικά, εν συγκρίση με προηγούμενες γενιέ ερευνητών στον τομέα. Αυτό το βλέπετε εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, στο γράφημα, απλό γράφημα, που δείχνει τις δύο βασικές παραμέτρους στον τομέα της ερευνάσμου. μου. Βλέπετε παρατήρηση του ουρανού, χρησιμοποιούμε τηλεσκόπια και πάμε μέχρι κάποιο βάθος. Όσο πιο βαθιά, στο διάστημα τόσο καλύτερα. Και το βλέπετε στο κάτω μέρος του διαγράμματος. Λοιπόν, η άλλη παράμετρος είναι η έκταση. Όσο μεγαλύτερη η έκταση του ουρανού που παρατηρείς, τόσο καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το διάγραμμα από αριστερά προς τα δεξιά ό,τι είναι δεξιά και κάτω στο διάγραμμα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα γκρίζα σύμβολα που βλέπετε εδώ είναι αποτελέσματα παλαιών ερευνών, παλαιά επιτεύγματα. Άρα πάνε στο πάνω αριστερό μέρος του διαγράμματος. Και τώρα τώρα με τη βελτίωση των οργάνων Έχουμε μεγαλύτερα σχέδια για το μέλλον, άρα μετά το 2020 θα έχουμε νέα μέσα και εργαλεία και θα καλυφθεί το κάτω δεξί τμήμα όπως θα προχωράμε. Και τα προγράμματα των οποίων ηγούμε με εξοπλισμό που θα έχει βελτιωθεί είναι στο μέσον μεταξύ του παρελθόντος και το μέλλοντος αυτό που κάνουμε τώρα. Κάνουμε άλματα πρόοδου, συνδέουμε παλιά έρευνα προετοιμάζοντας τις νέες έρευνες, τις μελλοντικές. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διαιρείται σε τρία τμήματα. Το πρώτο, ερευνούμε κάποιες πτυχές της αναπτύξεως των γαλαξιών και της συνιστώσεως αυτών. Μετά και η τρίτη πτυχή, η διασύνδεση όλων αυτών των πορισμάτων με τη μελλοντική έρευνα. Αρκετά για την αστροφυσική. να σας πω τι μου επέτρεψε να κάνω το ERC στην Κροατία. Το ERC λοιπόν μου έδωσε ευκαιρίες να δημιουργήσουμε τις πρώτες διεθνείς επιστημονικές ομάδες στην Κροατία, μία από τις ομάδες αυτές, που ασχολείται με την επιστήμη σε επίπεδο ανταγωνιστικό, υψηλό. Βλέπετε μια φωτογραφία της ομάδας. Έχουμε τρεις τρία PhD και τρία μεταδιδακτορικά διδακτορικά συγγνώμη, πτυχία. Και οι ερευνητές είναι από διάφορες χώρες για το με, μεταδιδακτορικό. Ο πρώτος ήταν τη Φιλανδία που είχε το διδακτορικό, ασχολείται με τα στοιχεία, επιστήμες δεδομένων στη Φιλανδία μετά από τρία χρόνια μαζί μας. Το δεύτερο μεταδιδακτορικό ε, από την Αυστραλία Εκείνη τελείωσε το συμβολό της πριν από μερικές εβδομάδες και πάει στην Νότια Αφρική για να εργαστεί στα πλαίσια ανεξάρτητης έρευνας μέσω υποτροφίας που πήρε και μια θέση. Και μετά είχαμε Ιταλό που πήρε την υποτροφία Μαρή Κιουρί και πάει στο Παρίσι για το μεταδιδακτορικό μέσω της ε, χορηγίας αυτής, μέσω της υποτροφίας Μαρή Curie. Υπέροχο τρόπο συνεργασίας, μια νέα ομάδα ερευνητών με καρποφόρα αποτελέσματα. Να τονίσω κάτι άλλο, ότι η χρηματοδότηση ERC μας επέτρεψε να έχουμε διεθνείς διασυνδέσεις. Χρησιμοποίησαμε αρκετά ποσά για να είμαστε δεμένοι με τους συνεργάτες σε διάφορες χώρες, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ και στην Χιλή, Φερρυπίνα. Ποια είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος. Δημοσιεύσαμε δημοσιεύματα που έχουν εξεταστεί από μοτίμους, περίπου 40 και πάνω από 15 ε, ε, συνετάχθησαν τα μέλη της στο Ζάγκρεπ. Έτσι μπορούσαν να εκπαιδευτούν έρευνητες που είναι πολύ επιτυχείς για να ε, ο πρώτο φοιτής που πήρε το PhD κάνει έρευνα στη Χαϊδελβέργη, στη Γερμανία, στο Ινστιτούτο Max ε, Planck με τα διδακτορικές έρευνε. Είχαμε και κάποια προσδόκητα αποτελέσματα. Τα μέσα στην ενημέρωση ε, ασχολήθηκαν με, τη, με τα χρήματα που διέθεσε το ERC. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, η ομάδα, ο διεθνής χαρακτήρας της ομάδας. Τελευταία 4-5 χρόνια προβλήθηκε σε, σε τηλεόραση, συνεντεύξει τηλεόραση, σε άθρα των εφημερίδων, γράψαν για μας. Μας δόθηκε δημοσιότητα, η οποία άνοιξε και διάβλο επικοινωνία προς το κοινό, περί επιστήμης, και αυτό είναι σημαντικό το το να απόψε. Thank you very much, Smolcic. Ευχαριστώ πολύ, Dr. Ε, Smolcic. Ακολουθεί ο Ισμαήλ Σεραλκεντίν, ιδρυτής, διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε ο τίτλος είναι «Έρευνα που ξεκινά από την περιέργεια». Εγώ πέρασα μέγα μέρος της ζωής μου στην Παγκόσμια Τράπεζα και συχνά μιλούσαμε με ανθρώπους και λέγαμε ότι ότι αν επενδύσουμε καλύτερα να φέρουμε αυτά που είναι ήδη στα εργαστήρια στην αγορά ή καλύτερα να επενδύσουμε στο ίδιο το εργαστήριο. Γιατί αυτό το δεύτερο μέρος χρειάζεται επίση στήριξη και καινοτομία. Θα ήταν όμως λάθος για θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση με την σημασία και την βαρύτητα που έχει να μην εξετάσουν και την έρευνα που βασίζεται στην περιέργεια και που έχει ουσιώδη σημασία γιατί έτσι ξεκινά η τεχνολογία. Και δεύτερο, δεν γνωρίζουμε που θα μας οδηγήσει, διότι ακριβώς η εφηρμοσμένη έρευνα εξετάζει πράγματα που είναι καταρχήν ήδη γνωστά. Η έρευνα εκ περιεργίας μας πηγαίνει πέρα από τα όρια. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει ε, να μεταμορφώσουμε τα πάντα, να στοχαστούμε λίγο τι έγινε πριν από 100 χρόνια περίπου όταν ένας άγνωστος εξάχρονος χωρίς διδακτορικό λεγόταν Einstein Albert το 1905 εξέδωσε πέντε μελέτες και άλλαξε τον κόσμο. Άλλοι μετά όπως ο μέγας επιστήμον Νίλς Μπορ άρχισε να δαπανά χρόνο προσπαθώντας να αντιληφθεί το πώς είναι φτιαγμένο το άτομο. Από εκεί ξεπίδησε η κβαντική φυσική και συνεχίστηκε. Είναι πολύ παράξενο. Δηλαδή είπαν κάποιοι τότε, μα σε τι μας σκεφτείτε αυτά. Όμως ολόκληρο το μισό του 20ου αιώνα με τα ηλεκτρονικά, τις επικοινωνίες από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν θα έχουν ξεκινήσει χωρίς αυτή την βάση. Όσοι λένε λοιπόν μη χάνετε το χρόνο σας με την έρευνα που βασίζεται στην περιέργεια θα είχαμε χάσει όλες τις εξελίξεις του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι να ρίξουν το βάρος τους στην έρευνα αυτή σημαντικό για όλους μας και σημαντικό να θυμηθεί κανείς επίσης ότι Βεβαίω και με τα 100, ίσω και περισσότερα, ελπίζω, δισεκατομμύρια ευρώ που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα αυτή, να μην ανοιχτεί μονάχα στην επιστήμη και η παγκόσμια επιστήμη κλπ. Αλλά να εξετάσουν και την σύγκληση μεταξύ των διαφορών επιστημονικών τομέων. Υπάρχει ένα τομέα την Bio-Info-Nanotechnology, την βιονανοτεχνολογία που μπορεί να ξεκινά από οτιδήποτε, από την καταχώρηση ε, μεγάλων όγκων δεδομένων μέχρι το DNA, ακόμα και τη συνθετική βιολογία. Δεύτερος τομέας που θα έλεγα να σκεφτείτε πολύ καλά είναι η πολυκλαδική ε, προσέγγιση περιβάλλον. Ε, διαφορές των φύλων, η κοινωνική, κοινωνικός αποκλεισμός και η κοινωνική συμπερίληψη. Και βεβαίως να ρίξετε ιδιαίτερο φως, να ρίξετε ιδιαίτερο βάρος στην Αφρική. Είναι 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι η Αφρική και μέχρι τέλους του αιώνα πάει να τετραπλασιαστεί. Λέει, λένε τα Ηνωμένα Έθνη Άλλοι λένε βέβαια, άλλοι φορεί λένε ότι θα τριπλασιαστεί. μιλάμε εδώ όμως για παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ενώ άλλε περιοχέ του κόσμου μειώνεται, μη βλέπουν να μειώνεται ο πληθυσμό τους. Γι' αυτό και θα γίνει πολύ δύσκολη η ζωή στην Αφρική. 95% της αγροτικής παραγωγής εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις. Επομένως οι γεωργοί δεν θα μπορούν να διατηρήσουν την ασφάλεια παροχή τροφίμων για ένα τέτοιο μεγάλο πληθυσμό και για τα αστικά κέντρα που αναπτύσσονται στην Ήπειρο αυτή. Ποιε θα είναι οι νέε πηγές ενέργειας, ε, τα εφιαστικά κέντρα κ.ο.κ. το Συνεργασία λοιπόν. Και εδώ έρχομαι στο τελευταίο. Πώς να συνεργαστούμε. Δυστυχώ στο παρελθόν υπήρχε η τάση να κάνουν ε, συνεργασία σε επίπεδο κυβερνήσεων, υπουργείων και ούτω εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προτείνει κάποιους τομείς που είναι προβληματικοί και να στοχεύσει σε αυτούς. Για παράδειγμα την ταξινόμηση της ε, βιολογικής, βιοποικιλότητας σε ορισμένε ε, χώρε ή περιοχέ του κόσμου. Και αυτό μπορεί να γίνει και σε ένα εργαστήριο στη Φιλανδία, για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι οι καθηγητέ και ερευνητέ στην Ευρώπη που θα χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη θα πρέπει να αναζητήσουν συνεργάτε στι ίδιε τι χώρε όπου θα διεξαχθεί η έρευνα. Και αυτοί θα διαλέξουν του καλύτερου συνεργάτε. Έτσι φτιάχνει κανεί πραγματική συνεργασία. Όταν επιστήμονε και ερευνητέ συνέρχονται για να επιλύσουν κοινά προβλήματα, όπω του παγκοσμίου κλίματος αντί να προσπαθούν να διοχετεύσουν τις προσπάθειες αυτές μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες, Υπουργείο και το καθεξής. Έχοντας πει αυτά, θεωρώ ότι θα έχουμε πολλές δυνατότητες να μεγιστοποιήσουμε την χρήση της τεράστιας αυτής ευκαιρίας που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαραγγελντίν. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζούλη Μάξ, την εκταλιστική διευθύντρια από τη Royal Society του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ πολύ, Jean Πιέρ Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοτσιγιώμη, Όμισαν, για την ε, συμβολή σας και για την έμπνευση και το όραμα που δημιουργήσατε αυτό το STS Forum στο Κιώτο. Η Royal Society, η Βασιλική Εταιρεία, είναι η Εθνική Ακαδημία Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει ε, εδώ και 350 χρόνια. Από την αρχή όμως είχε διεθνές ε, ενδιαφέρον ε, εκεί είχε στραμμένο δηλαδή το ενδιαφέρον της. Ε, αρχικά ε, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν σε εξερευνητικές αποστολές στην Αρκτική, νωρίτερα σε άλλες υπήρους είχαμε τους εξερευνητές. Τώρα έχουμε την αρχική αποστολή που είναι η πρόθεση της αριστείας στην επιστήμη. Στηρίζουμε την επιστήμη αναγνωρίζουμε από την ευρύτερη δυνατή έννοια την καλύτερη επιστήμη όπου και αυτή αν πραγματοποιείται στον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι η Βασιλική Εταιρεία εργάζεται με πάνω από 60 χώρες ε, στον κόσμο, εκ των οποίων ορισμένες έχουν ε, έρευνα, ε, την καλύτερη έρευνα που, που κινείται από την περιέργεια, άλλη εφαρμοσμένη έρευνα δεν φυσικά άλλοι αποκλείεται το ένα από το άλλο. Άλλοι επιστήμονες, μάλλον σε άλλες χώρες, είναι στα σπάργανα ακόμη εκεί η επιστήμη και κάνουμε πολλή δουλειά. Για να πιάσω μετά από αυτό που είπε Ισμέλ για την Αφρική, εμείς θα ξεκινήσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στην Αφρική, πάνω από 20 χρόνια εργαζόμαστε στην Αφρική, αλλά τώρα θα επεξεργαστούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα, ένα project για τους ε, μελλοντικού ηγέτες ε, της Αφρικής στον τομέα των επιστημών. Έρχομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το Horizon Ευρώπη είναι μια φανταστική ευκαιρία. Το επίπεδο του προπλησμού είναι καταπληκτικό. Μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια. Καταπληκτικό. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπήρξαν πολλές ενδείξεις που οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη κοιτάζει πέρα από την Ευρώπη, κοιτάζει τη θέση που έχει στην παγκόσμια σκαγκέρα. Και στην έκθεση Λαμή που αναφέρθηκε κατά το, στις προηγούμενες συνεδρίες, Lab Fab app είναι τα συντετμημένα της, ε, το συντετμένο όνομα έχει μεγάλη, δίνει μεγάλη σημασία ε, στην ε, έρευνα κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε έναν κόσμο που με όλο και περισσότερο και η επιτυχία βασίζεται στην παραγωγή, τη μετατροπή, γνώση και Αυτά τα λέει αυτή η έκθεση και λέει ότι η ε, συνεργασία είναι, αν θέλετε, το σήμα κατά τεθέν ε, της ε, έρευνα και καινοτομία. Δηλαδή, αυτός ο πολύ σημαντικός φορέας που προσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να είναι πραγματικοί ηγέτες μέσω και του προγράμματος Horizon Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο και τα σχετικά προγράμματα είναι προγράμματα κατ' ουσίαν, δηλαδή δίνουν ευκαιρίες συνεργασίας με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να είναι κοντά ή μακριά γεωγραφικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκουν εδώ εκπρόσωποι και ε, από τις δύο κατηγορίες χωρών. Προωθείται λοιπόν ε, και η εφαρμοσμένη στις επιστήμες αλλά και η ε, έρευνα που βασίζεται στην περι... και υποκίνητα από την περιέργεια. Ανανεωμένη στο ε, θεματολόγιο για την έρευνα, την καινοτομία, η ευκαιρία της Ευρώπης για χάραξη και διαμόρφωση του μέλλοντος, όχι του μελλοντοστής, του μέλλοντος. Αυτό είναι ένα έγγραφο, μια ανακοίνωση της Κομισιόν, μου την προηγούμενη εβδομάδα και είναι σημαντικό. Επίσης νωρίτερα έγινε λόγος για τις επενδύσεις που κάνει η Ιαπωνία ε, στην έρευνα και καινοτομία. 1,3% του ΑΕΠ βάζει η Ευρώπη. Η Ιαπωνία 2,6%. Το διπλάσιο δηλαδή από την ε, πλευρά ε, των επιχειρήσεων. Νομίζω όμως ότι αναφέρθηκαν ορισμένοι σε αυτό το νέο έγγραφο για τα venture capital που μιλά για την επιστήμη και την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν όλες τις επιτυχίες ε, για να υπάρξουν ε, ε, νέα επιτεύγματα και να αλλάξουν τα παραδείγματα και τα μοντέλα για μια νέα ευημερία προς όφελος της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ. Thank Και τώρα να δώσω το λόγο στον Δόκτωρ Μότ Κοκοτάνη, θελεστικό διευθυντή του Weekend Japan σου και είναι μαθηματικός. Μοτόκο. Η κυρία Κοτάνη. Ευχαριστώ. Μεγάλη χαρά για μένα να παρίσταμε, να μοιραστώ μαζί μας, μαζί σας τις ιδέες μου. Πώς στηρίζεται η έρευνα που βασίζεται στην περιέργεια. Λοιπόν, είναι παγκόσμια ε, η τάση αυτή όπου η έρευνα οδηγεί στην καινοτομία. Μιλείς μόνο όμως ότι βασίζεται στις ώρες γνώσεων μέσω έρευνας που διεξάγεται με βάση την περιέργεια. Είμαι μαθηματικός. Τα μαθηματικά συχνά είναι η γλώσσα του σύμπαντος και όλου του κόσμου και συνέβαλε στην ανάπτυξη επιστημών και, ε, και τεχνολογίας μέσω το πλαίσιο μαθηματικές έννοιες, οι σειρές, οι τύποι, ήταν έμπνευση στον επιστημονικό τομέα. Και οι μαθηματικοί μπόρεσαν να αναπτύξουν και νέα μαθηματικά με την εξέλιξη. Πρόσφατα, η εποχή των μαθηματικών ήταν μια έκθεση που βγήκε στον Ηνωμένο Βασίλειο και αναφέρθηκε στην ανάγκη για, για εταιρείε, για ένωση, για νέα μαθηματικά δεδομένα. και πώς σχετίζεται με την έρευνα. Και βάσει των μαθηματικών ιδεών ε, να προχωρήσουμε που αναπτύχθηκαν κατά το παρελθόν. Παράδειγμα, η αριθμητική σειρά είναι στην καρδιά των μαθηματικών. Η αριθμητική σειρά είναι όμορφη. θα ακούσατε μια ιδέα που αναφέρθηκε το 1637 που αφορούσε τη σειρά, άρα χρονολογείται από 360 χρόνια. Α, και διατυπώσανε οι Ιάπωνες μαθηματικοί την ερώτηση για την εθνική σειρά, βήσαν τη σχέση που υπήρχε μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που είχαν. αλλά την αριθμητική σειρά δεν μπορούσαν να την εμφαρμόσουν ε, την ιδέα αυτή στην πρακτική. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Τώρα όμως είναι κλειδί στην κρυπτογράφηση δεδομένων για την ασφάλεια των δεδομένων στις επικοινωνίες. Πολύ σημαντική αυτή η κρυπτογράφηση για την ψηφιακή κοινωνία. Το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε πριν από 100 χρόνια και η ύπαρξη του Πανεπιστημίου ήταν βασικό στοιχείο για την εθνική στρατηγική και άλλαξε δραματικά την Ιαπωνική βιομηχανία. Κάποιοι είχαν ελευθερία οι Ιάπωνες ερευνητές να ικανοποιήσουν τη δίψα τους για την έρευνα και την περιεργία τους. Αυτό έδωσε άριστα αποτελέσματα ερευνητικά. Το βλέπουμε τις επιτυχίες. Από το Νόμπελ που, ανατέθ, που απενεμήθη στην Ιαπωνία. Η καινοτομία η έρευνα και η καινοτομία και η έρευνα που ασύστη στην περιέργεια, όλα αυτά ενέπνευσαν το ένα το άλλο και εξελίσσονται. Όπως εξήγησα. Εκπροσωπώ το Ρίκεν. Να μιλήσω για το Ρίκεν. Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τις Φυσικές Επιστήμες. Είναι παράδεισο των επιστημόνων. Το λέμε αυτό όχι γιατί παίρνουν πολλά χρήματα οι ερευνητέ, αλλά έχουν μεγάλη ελευθερία για να κάνουν έρευνα με βάση την περιέργειά του. Το Ρίκεν παρουσίασε τη δική του, παράγει έρευνα παγκόσμια ε, κλάση. Έχει και έξοχες υποδομές που παρέχει στους Ιάπωνες ερευνητές και στον υπόλοιπο κόσμο. Σημαντικότατο να υπάρχει αυτή η υποδομή για ευρεία χρήση. Το Πανεπιστήμιο Μανάκα βρήκε κάποια κύτταρα που ήταν ε, ε, έκανε μεγάλη πρόοδο στον τομέα της έρευνας που αφορά τους ιούς. Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων και δεδομένα. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε δεν είχε σαν στόχο να βρει το, το κύτταρο IP, αλλά ήταν ευρέως διαδεδομε... χρησιμοποιημένη βάση δεδομένων. Και το Ρίκεν έκανε κλινικές δοκιμές για ε, την ιατρική στο τομέα της αναγέννησης των κυτάρων. και βοηθάει αυτού του είδους υποστήριξη και υποδομές στο να γίνονται ρηξικέλευτες ανακαλύψεις. Το νέο πλαίσιο του ορίζοντας Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί είπαν ότι η διεθνή συνεργασία είναι σημαντικότατη. Το Ρίκεν είναι μικρός φορέας. Στηρίζουμε όμως την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ενώσης Ιαπωνίας. Ο διευθυντής είπε ότι το Ρίκεν θα ανοίξει γραφείο στις Βρυξέλλες τον Αύγουστο, το φθινόπωρο, θα είναι ευρωπαϊκό γραφείο, με τα χαράς να συνεργαστούμε για την έρευνα βάση της περιέργειας και να προχωρήσουμε στην καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. I think for... Μας μένουν λίγα λεπτά για ερωτήσεις αν έχετε να υποβάλλετε γιατί είμαστε βέβαια πάλι εντός των ορίων του χρόνου μας λόγω της ε, πραγματικά θαυμάσιας ε, θαυμάσιου χειρισμού του χρόνου από τους ε, ομιλητές μας. Έχετε παρακαλώ ερωτήσεις. Όχι, καλώς, δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Τότε θα παρακαλέσω τον πρόεδρο Όμη να έλθει εδώ στο έδρανο, αφού ευχαριστήσω και πάλι τις ομιλήτριες, μπορούν να επιστρέψουν αν θέλουν στις θέσεις των.

Αγαπητέ Συμπρόεδρε, έγιναν δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων. Ήρθε όμως πια η ώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή. Όταν ήρθα, είδα ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα. Το πρόγραμμα για τη Βόρεια Κορέα, με τη συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείες, για την ε, Μέση Ανατολή. Είδαμε ότι υπάρχουν και πολλά προγράμματα ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουμε το μέλλον. Αλλά ε, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες του μέλλοντος το μέλλον της ανθρωπότητας. Βέβαια έχουμε πολλά προβλήματα να επιλύσουμε τα επόμενα χρόνια. Θα θέλαμε πολύ να επαναληφθεί η συνάντηση αυτή με τις χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου. Βεβαίως γνωρίζω ότι υπάρχουν οι ευρωεκλογέ, προβλέπονται οι ευρωεκλογέ την επόμενη χρονιά. Όμως η επιστήμη και η τεχνολογία θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και θα είναι βεβαίως η πόρτα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Ας καθίσουμε μαζί όλοι γύρω από ένα τραπέζι να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Ο πρόεδρος Μπουργκινιό. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Αντιλαμβάνεστε ότι η παρούσα συνεδρία ήταν κοινή μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών, αν και εγώ δεν είμαι ευρωβουλευτή. Παρ' όλα αυτά ευχαριστώ τις δύο επιτροπές, Επιτροπή, επιτροπή ε, αλλά και τη ΣΤΟΑ που γνωρίζετε δεν είναι κοινοβουλευτική επιτροπή, είναι επιτροπή μεν, αλλά ασχολείται με την αξιολόγηση τεχνολογία. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνωμονε για την φιλοξενία του και βεβαίω το Science in Society Forum είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει ο πρόεδρος Όμι. Σας λέγω ότι πρόκειται για μια εξαιρετική θαυμάσια πλατφόρμα για ανταλλαγές απόψεων μεταξύ επιστημόνων, ερευνητών, επιχειρηματιών, ανθρώπων που λαμβάνουν τις αποφάσεις στο πολιτικό επίπεδο. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας είναι λοιπόν σημαντική και μου ανετέθη να μεταφέρω τις ευχαριστίες του Προέδρου ε, Καθηγητού και πρώην Υπουργού κυρίου Μπούσεκ και του Δ. Ρούμπικ ε, ε, τις ευχαριστίες λοιπόν για την συνάντηση αυτή. Το επόμενο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των δύο πάνελ για τις παρεμβάσεις τους και ιδίως διότι φώτισαν το θέμα της διεθνούς συνεργασίας από διάφορες πλευρές και για το πώς τεχνολογία και καινοτομία μπορούν να συνδυαστούν. Βεβαίω και όλου του ευρωβουλευτέ που συμμετείχαν και που έθεσαν ερωτήσει. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε και στον Επίτροπο κ. Μοέντα που προσήλθε και ε, συνέβαλε στην ε, επιτυχή διεξαγωγή της συνεδρίασης με σημαντικέ παρεμβάσει και επειδή βρισκόμαστε στη σημαντική φάση τη προετοιμασία του προγράμματο Horizon Ευρώπη και το έγγραφο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι διαθέσιμο πλέον στις 6-7 έκτου. Πολύ σύντομα δηλαδή. Κάτι που έχει ήδη επιτευχθεί, έχει διασφαλιστεί, είναι τα χρήματα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αποθεματικό το μαγικό νούμερο, μαγικό αριθμός των 100 δισεκατομμυρίων που προβλέπει ο κ. Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα αυτό, ε, ήταν αποτέλεσμα σημαντικού αγώνα. Ακούσατε επίση ότι από την πλευρά του Κοινοβουλίου εκφράζουν μεν την ικανοποίησή τους για τα 100 δισεκατομμύρια. Ελπίζουν ωστόσο θα μπορέσουν να τα αυξήσουν, να φτάσουν μέχρι και τα 120, δηλαδή να το διπλασιάσουν όπως είχε ε, ζητηθεί και από την ομάδα Λαμή. Ε, έχουμε λοιπόν μεγάλες προσδοκίες για την τελική φάση του Horizon Europe που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις όπως συμβαίνει πάντοτε στην Ευρώπη ε, ξεκινώντας από την πρόταση Επιτροπής, συζήτηση στο Κοινοβούλιο και συζήτηση στο και με το Συμβούλιο, δηλαδή στους προσώπους των χωρών μελών. Ελπίζω οι συζητήσεις αυτές να αποδειχθούν αποτελεσματικές και επειδή είμαι και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και όχι επίτροπος, ελπίζω το πρόγραμμα και το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνών ε, να αποδειχθεί σημαντικό. Πιστεύουμε στη συνέχεια, διότι θεωρούμε το πρόγραμμα είναι σημαντικό και πρέπει η δομή του να διατηρηθεί και οι ευθύνε αντίθεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Δεύτερον, κινητικότητα, agility. Ορισμένα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, δηλαδή καλύτερη παρακολούθηση των επιπτώσεων του προγράμματο. Και το τρίτο είναι διεθνή συνεργασία πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα και αυτή για την οποία θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε ε, ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες και το τέλος αύξηση της κλίμακας δηλαδή αύξηση του προϋπολογισμού. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους Ιάπωνες συναδέλφους για τη θαυμάσια συνεργασία. Προσωπικά έχω επισκεφθεί κατ' επανάληψη την Ιαπωνία και έχω συνεργαστεί με εκπροσώπους πολλών φορέων στην Ιαπωνία και πάντοτε θεώρησα ότι ήταν ε, ε, τεράστιο το όφελος από, την, ε, από τις επαφές αυτές κάτι που ακούσατε ήδη κατ' επανάληψη και ίσως πρέπει να το διδαχθούν και οι Ευρωπαίοι και το ανέφερε και ο Δόκτωρ Ρούμπικ είναι η πολύ μεγάλη σημασία που αποδίδουν οι Ιάπωνες στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πέτο μου έχω και το σύμβολο των στόχων αυτών και για μένα είναι σημαντικό σημάδι ότι η Ιαπωνία εντάσσει στην πολιτική ερευνών της στους στόχους αυτούς. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ καλός ιονός αυτός και ελπίζω να τον αντιγράψουν και άλλοι. Αντιλαμβάνεστε ότι θεωρώ δυστυχώς ότι κάποιοι δεν το πράττουν. Τέλος για τη διεθνή συνεργασία, μόλις επέστρεψα από τη Μόσχα σήμερα το πρωί και θα ήθελα να σας ε, πω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι η επιστημονική διπλωματία είναι πάρα πολύ σημαντική παρόλο που υπάρχουν εντάσεις μεταξύ της ρωσικής κυβερνήσεως. Βέβαια, οι Ρώσοι επιστήμονες θέλουν να συνεργαστούν, θεωρούν ότι η επιστήμη πάντοτε μπορεί να δώσει χώρο για συζήτηση, για ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων και ακούσαμε και χθε το βράδυ ξεκάθαρα λόγια ανοίγματο προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τη συμμετοχή σας σήμερα το απόγευμα. Ελπίζω να ωφεληθήκατε από τις απόψεις που ακούστηκαν και από τα θέματα που συζητήθηκαν. Θα βρείτε αναψυκτικά και μια δυνατότητα επαφών εκτός της αιθούσης. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.